Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Ε, είναι υπερπλήρες ε, το πρόγραμμα το διήμερο της Επιτροπής Βιομηχανίας. Δυστυχώς ο πρόεδρος μας σήμερα κολλείται και δεν μπορεί να προεδρεύσει οπότε θα προεδρεύσει ο υποφαινόμενος. Έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχατε λάβει. Οπότε να σας παρουσιάσω την σημερινή και αυριανή μέρη σε διάταξη. Σήμερα, μετά το πέρας της ακρόασης, θα συζητήσουμε το σημείο 7 δηλαδή την ενημέρωση για την αποστολή της ήτρε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. Και το σημείο 6 του αρχικού σχεδίου έγκρισης, δηλαδή συμφωνία με τη Βραζιλία, θα αναβληθεί για αύριο, για την αυριανή συνεδρίαση που θα συζητηθεί στο τέλος. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να την εγκρίνουμε με τις προτινόμενες αλλαγές. Συμφωνείτε? Μήπως υπάρχουν σχόλια? Όχι. Οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Περνάμε στη δημόσια κρόση τώρα για το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για την πράξη για την κυβερνοασφάλεια. Cyber Security Act. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους τέσσερις καλεσμένους μας ε, θα χωρίσουμε σε δύο ενότητες ε, την ακρόαση. Στην πρώτη ενότητα θα ακούσουμε τους πρώτους δύο καλεσμένους, τον κύριο Σάμπα Χιούζερ και την κυρία Μόιρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους καλεσμένους μας ομιλητές ε, να τηρήσουν τους συνήθεις δηλαδή γύρω στα 8 λεπτά για τις αρχικές τους παρουσιάσεις. Κατόπιν θα ακούσουμε τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές που θα έχουν την ευκαιρία να εκφέρουν τη γνώμη τους μέσα σε δύο λεπτά και στη συνέχεια συζήτηση με την ομίγυρη ε, με ομιλητές βουλευτές για ένα λεπτό στον καθένα. Για το θέμα αυτό τη πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε τη σχετική πρόταση κανονισμού για την πράξη της κυβερνοασφάλειας στι 13 Σεπτεμβρίου του 2017. Ο κανονισμός απαρτίζεται από δύο σκέλη. Το πρώτο προβλέπει μια διεύρυνση και αναβάθμιση της εντολής του Οργανισμού για την ε, Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και δεύτερο σκέλος, ένα προαιρετικό σύστημα για την πιστοποίηση για θέματα κυβερνοασφάλειας. Εμείς, η Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας, είμαστε κατ' ουσία αρμόδια επιτροπή. Οι συζητήσεις βέβαια περί αρμοδιοτήτων συνεχίζονται, οπότε θα ήθελα να καλωσορίσω το, την εισηγήτρια της Επιτροπής μας, την κυρία Αντζέλικα Νίμπλερ. Δεν τη βλέπω βέβαια στην αίθουσα. Ελπίζω όμως ότι θα έρθει εντωμεταξύ και τον κύριο Γιάνν Φιλίπ Άλμπρεχτ που αντικαθιστά τον συντάκτη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τη ΣΥΜΚΟ. Ελπίζω να έρθει και ο κύριος Άλμπρεχτ σε λίγο. Έχουμε και τον εκπρόσωπο, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Δέσποινα Σπανού, που είναι Διευθύντρια για την Ψηφιακή Κοινωνία, την Εμπιστοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, του ΕΝΙΣΑ. Ε, ο κύριος Πέρσερ είναι ο εκπρόσωπος του ΕΝΙΣΑ, που είναι τμήματάρχης ε, στις ε, βασικές λειτουργίες. Κατά πάση πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει, θα αναγγείλει την πρότασή της για την πράξη κυβερνοασφάλειας στις 23 Ιανουαρίου του 2018. Όπως είπα και προηγουμένως, θα διαιρέσουμε την ακρόαση σε δύο τμήματα και μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις θα έχετε όλη την ευκαιρία να θέσετε τις ερωτήσεις σας ή να κάνετε δηλώσεις. Το πρώτο, το πρώτο τμήμα της ακρόασης προβλέπει τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τον Οργανισμό ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, τον ΕΝΙΣΑ. Θα δώσω το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Γκέρχαρτ Σάπχουζερ, που είναι αντιπρόεδρο του Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Ασφάλεια των Πληροφοριών. Ο κύριο Σάπχουζερ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στη θέση του Αντιπροέδρου του Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Ασφάλεια των Πληροφοριών την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτου. Αποφύτησε με πτυχίο μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ και κατόπιν ε, έλαβε ε, διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ στο Πανεπιστήμιο της Χάγης. Το Νοέμβριο του 1991 προσχώρησε στο Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, το BSI στα γερμανικά, και εδώ και 26 χρόνια εργάζεται σε αυτό το ομοσπονδιακό γραφείο. Είναι εμπειρογνώμονας ειδικό σε θέματα κρυπτογράφησης, ασφάλειας των πληροφοριών, εφαρμογής και εποπτείας. Μετά την παρουσίασή του, μετά τη σύντομη παρουσίαση που σας έκανα του καλεσμένου μας, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαπχιούζερ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρία Μόγκερ, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που ε, έχω την ευκαιρία να σας απευθύνω τον λόγο σήμερα. Μιλούμε για το Cyber Security Act, την νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια και για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου πιστοποίησης για το ΕΝΙΣΑ. Η Γερμανία έχει υποστηρίξει εξ αρχής την δημιουργία του ΕΝΙΣΑ από το 2004 και έχει συμβάλει στην δημιουργία του οργανισμού αυτού. Έχει δε εποφεληθεί από την εργασία του οργανισμού αυτού, όπως και αυτός ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ δηλαδή, έχει εποφεληθεί από την εργασία του οργανικού μας οργανισμού BSI. E, σε ένα τρόπο αλληλοϊποστηρικτικό ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κύβερνο ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ανταποκρίνεται και στην ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Η κεντρική αποστολή του Ένισα για μας είναι να είναι βασικός αρμόδιος συνομιλητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε τι που έχει σχέση με την ασφάλεια δικτύων, δηλαδή Key Point of Reference στα αγγλικά. Και εννοώ με αυτό την διάθεση εμπειρογνωμοσύνης και παροχή συμβουλών για θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφορικής υποστήριξη προς τις χώρες μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη δημιουργία ικανοτήτων NIS, καθώς και στήριξη που προσφέρει για την νομοθετική διαδικασία. Η προώθηση πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ όλων των stakeholders στα NIS, δηλαδή παράδειγμα με την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ο οργανισμός ενίσα λόγω της σημασίας της ασφάλειας των δικτύων και της πληροφορικής δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με την νυν μορφή του. Το έτος 2017 είδε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κρίσεις κυβερνοασφάλειας που οδήγησαν την κοινωνία, τα κράτη και την πολιτική γενικότερα να αντι, αντιληφθούν τη σημασία του θέματος. Και βεβαίως καθώς προχωρεί η ψηφιοποίηση της κοινωνίας, στο μέλλον τα πράγματα αυτά θα γίνουν όλο και σημαντικότερα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο κανονισμό ένισα σωστά προβλέπει και ζητεί διαρκή εντολή για τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ, κάτι το οποίο χαιρετίζουμε απολύτως εμείς από γερμανική πλευρά. Υποστηρίζουμε επίσης ως Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την αύξηση των πόρων του ΕΝΙΣΑ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντά του. Τονίζουμε επίσης τη σημασία του ΕΝΙΣΑ για την εφαρμογή της οδηγίας NIS από το έτος 2016 και σημαντική βέβαια, σημαντικό μάλλον ρόλο αναλαμβάνει στα όργανα προβλέπονται στην οδηγία εκείνη, δηλαδή την ομάδα συνεργασίας και το δίκτυο της ομάδας για την αντιμετώπιση επεισοδίων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η αξιολόγηση του έργου του Έλισσα είναι θετική για, για μας από γερμανικής πλευράς, διότι ήδη έχει προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στις χώρες μέλη. Θυμίζω για παράδειγμα την επεξεργασία συστάσεων για την επέκταση εθνικών CSIRT, δηλαδή ομάδων για την αντιμετώπιση επεισοδίων υπολογιστών, το Cyber Europe, πανευρωπαϊκές ασκήσεις, πολύ σημαντικό θέμα, ή και την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Μήνα Κύβερνο Ασφάλειας, European Cyber Security Month, δηλαδή παροχή πληροφοριών, ευαισθητοποίηση και ούτω Ο νόμος περί κυβερνοασφάλειας που συζητείτε σήμερα εσείς αποδίδει την σημασία του ρόλου του ένισα. Όμως η πρόταση την οποία συζητείτε περιλαμβάνει και ορισμένα, ορισμένες νέες έντολες, νέα καθήκοντα για τον οργανισμό. Δηλαδή ε, προβλέπει έναν ρόλο για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Στην πρόταση που συζητείτε, ο ρόλος που προβλέπεται για τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ, κατά τη γνώμη μας, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη δραστηριότητα πιστοποίησης των χωρών μελών, όπως αυτή ασκείται σήμερα, και την επιτυχή συνεργασία με τη βιομηχανία, η οποία μάλιστα αναγνωρίζεται και διεθνώς και πέραν δηλαδή των ορίων της Ευρώπης. Για να εφαρμοστεί το πλαίσιο πιστοποίησης με την προτινόμενη μορφή, αυτό ενδέχεται να αποδυναμώσει την πιστοποιητική δραστηριότητα των χωρών μελών και να μειώσει το επίπεδο, του, το επίπεδο ασφαλείας λόγω της διαρκούς προόδου της ψηφιοποίησης αλλά και της εντάσσεως των κινδύνων θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα έχει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για αυτό το θέμα θα τοποθετηθούμε ως BSE και στην επόμενη φάση της ακροάσεως. Εξάλλου η νέα πρόταση εντολής προβλέπει νέο ρόλο του ΕΝΙΣΑ για την επιχειρησιακή συνεργασία, δηλαδή αύξηση του ρόλου στην συνεργασία για την αντιμετώπιση κυβερνοκρίσεων. Ανάλυση, αναλυτική ικανότητα για την αντιμετώπιση επεισοδίων με σημαντικές ε, επιπτώσεις εφόσον το ζητήσει μια χώρα μέλος. Εμείς ως Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την πρόταση για αύξηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του οργανισμού ένισα και οι λόγοι που μα παρακινούν σε αυτή την επιφυλακτικότητα είναι η εξή. Αφενό θεωρούμε την κυβερνοασφάλεια ω κυρίω εθνική αρμοδιότητα. Λόγω τη κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών μελών, και χωρών μελών αλλά και του ΝΑΤΟ δευτερευόντω, αλλά και λόγω τη αρχή τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα, οι βασικέ αρμοδιότητε κυβερνοασφάλειας ανατίθεται στι χώρε μέλη. Η μετατόπιση αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσει στην μείωση των προσπαθειών των χωρών μελών για την αύξηση της κυβερνοασφάλειας. Από τη δική μας εμπειρία, άλλωστε, γνωρίζουμε ότι σε κανένα άλλο τομέα δεν είναι τόσο σημαντική η εμπιστοσύνη των εθνικών φορέων όπως στον τομέα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εμπιστοσύνη στους εθνικούς οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν λεπτομερή γνώση και εγκύτητα στις ομάδες στόχους, είτε πρόκειται για τη δημόσια διοίκηση, για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις κρίσιμες υποδομές, οι οποίες σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για ένα επίπεδο εμπιστοσύνη το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από συνεργασία πολλών ετών. Δεύτερο, υπάρχουν ήδη φορείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι επιχειρησιακά λειτουργικοί. Υπάρχει στο επίπεδο της ομάδας αντιμετώπισης επεισοδίων ηλεκτρονικών υπολογιστών, το CERT-EU, το οποίο έχει την αρμοδιότητα χωρίς πιστοποίησεων και βεβαίω υποφελείται από την ροή πληροφοριών από όλε τι χώρε μέλη. Το CRTU είναι ευρωπαϊκό επιχειρησιακό φορέα και είναι σε θέση λοιπόν στον δικό του χώρο αρμοδιοτήτων, που είναι τα ευρωπαϊκά όργανα και ευρωπαϊκέ αρχέ, να χορηγεί τι αναγκαίε πληροφορίε. Δηλαδή να εξηγεί ποια είναι η κατάσταση και να προσφέρει και υποστήριξη για την αντιμετώπιση επεισοδιών. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κυβερνοκρίσεων, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται κυρίως για κρίσεις εθνικού χαρακτήρα με μια ευρωπαϊκή διάσταση. Η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να αρθεί ειδικά για τον κυβερνοχώρο. Μπορεί να προκύψει προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια μέσω του ένισα μόνο εφόσον βασίζεται στη συνεργασία των χωρών μελών και μάλιστα να ξεπερνά το επίπεδο αυτό. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κρίσεις κυβερνοασφάλειας που να ανατεθεί σε μια ευρωπαϊκή αρχή, κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται να εντείνει την εμπιστοσύνη των δικτύων. Κυρίως εθνικές δομές, οι οποίες λειτουργούν ήδη και οι υφιστάμενες ικανότητες σε όλες τις χώρες μέλη αποτελούν την βάση για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ιδίω η δεσμευτική ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών καθώς και η διεύρυνση, η αύξηση των ειδικών φορέων και οργανισμών με επιχειρησιακή ικανότητα είναι σημαντικές για την αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι μια common situational awareness στο επίπεδο των χωρών μελών για να μπορούν να αντιμετωπίζονται ή δυνατόν να συντομεύεται, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω με ένα συμπέρασμα, το οποίο συμπέρασμα έχει ως εξής. Θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε πρώτα-πρώτα το εφικτό, την εφικτότητα δηλαδή, και την αποτελεσματικότητα, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι προτιμότερη μια συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών παρά ανάθεση επιπλέον καθηκόντων σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό οργανισμό που εν τέλει θα οδηγήσει σε προσδοκίες οι οποίες δεν θα μπορούν να εκπληρωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σα για απάντηση ερωτήσεων. Ευχαριστώ κύριε Σαπ Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας. Θα μπορούσατε, είμαι βέβαιος, να μιλήσετε πολλές ώρες για το θέμα αυτό. Είστε άλλωστε ε, ε, εμπειρογνώμων, είστε ειδικό στο θέμα αυτό. Αλλά δυστυχώς υπάρχει κάποια πίεση χρόνου. Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάντως και πάλι. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Μόγκρα, που είναι διευθύντρια στο κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ για την συνεργάσιμη κυβερνοάμυνα. Το υπόβαθρο της κυρίας Μόγκρε ε, ήταν ε, υποδιευθύντρια στο γραφείο επαφής του ΝΑΤΟ στο ΚΙΕΦ. Ε, έχει αναλάβει στο κέντρο από το Σεπτέμβριο του 2017. Προηγουμένως ήταν ε, σύμβουλος για θέματα πολιτικής ασφάλειας στο, ε, παρά το πρόεδρο της Εστονίας 2012 με 2017 και επίσης ε, υπηρέτησε ως ε, υποδιευθύντρια στο γραφείο του ΝΑΤΟ στο Κίεβο και στο τμήμα για το ΝΑΤΟ του Εστονικού Υπουργείου Άμυνας για την προώθηση της προσχώρησης της χώρας της στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα έχει πτυχία από το King's College, από το Middleburg College και από το Πανεπιστήμιο του Ταρτού. Σπούδασε και στο κέντρο της Μπολόνια, του Johns Hopkins Science και επίσης στο Παρισινό Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών της ε, Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ήτρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα σας μιλήσω ως ανεξάρτητη εξωτερική εμπειρογνώμων. Είμαι πρόεδρος ε, του Κέντρου ε, Αριστείας του ΝΑΤΟ για την συνεργάσιμη με κυβερνοάμυνα. Πρόκειται για ένα και το που βρίσκεται στο Τάλιν της Εστονίας και ήμουν και πρώην ε, σύμβουλος για θέματα ασφαλείας ε, στον πρόεδρο της Εστονίας. Στο κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ, στο κέντρο μας, ε, έχουμε ένα μείγμα, ποικιλόμορφο μείγμα εμπειρογνωμόνων από το στρατό, τις κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια, τον κλάδο που συνεργάζονται στο κέντρο μας. Επικεντρωνόμαστε σε έρευνα, ε, κατάρτιση και ασκήσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς. Ε, την τεχνολογία, τη στρατηγική, ε, τη σχετική νομοθεσία και τις κυρώσεις. Και μάλιστα δίνουμε μια πολύ συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη σκοπιά για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. θα σας δώσω από πρώτο χέρι εμπειρίες για να σας πω ότι κατά τη γνώμη μας είναι κρίσιμο για θέματα αυτά προκειμένου να δημιουργήσουμε την αθεκτικότητα και των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι, ότι ο αριθμός και η πολυμορφία των κυβερνοαπειλών αυξάνονται. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την αθεκτικότητά της στις κυβερνοεπιθέσεις. Με Μέσω της νέας εντολής, ο, ο υφιστάμενος ρόλος του ΕΝΙΣΑ θα ενισχυθεί σε θέματα συνεργασίας για τις κυβερνοκρίσεις, διαχείριση των κυβερνοκρίσεων και προστασία των κρίσιμων υποδομών. Μάλιστα ήδη ο ΕΝΗΣΑ εξασφάλισε προστιθέμενη αξία για τα θέματα αυτά, γιατί από το 2010 έχει αναλάβει την ευθύνη για την οργάνωση των πανευρωπαϊκών ασκήσεων με τίτλο «Κυβερνοευρώπη». Και τώρα θα σας μιλήσω από την εμπειρία που έχουμε από πρώτο χέρι και ως Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας του ΝΑΤΟ και ως πρώην σύμβουλος για θέματα ασφαλείας ε, του Προέδρου της Εστονίας. Πιστεύω ότι οι ασκήσεις στα γυμνάσια είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσουμε ικανότητες και να φτιάξουμε δεξιότητες. Η σημασία των ασκήσεων κυβερνοασφάλειας ε, είναι δεδομένη και απολύτως απαραίτητη για να, για να αντιμετωπιστούν κάποιες ε, ε, στρατηγικές απειλές που ε, γύρονται λόγω των κυβερνοκρίσεων. Επίσης ε, θέλουμε κατευθυντήρες γραμμές για να αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα παρόμοιες κρίσεις. Και μάλιστα υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και κάθε χρόνο οργανώνουμε ή βοηθούμε στην οργάνωση ασκήσεων του, του κυβερνοσυνασπισμού και τα Lock που κατά τη γνώμη μας είναι οι μεγαλύτερη εμβέλειας ασκήσεις για την κυβερνοασφάλεια. Και από το 2010 ε, ασχοληθήκαμε με την κατάρτιση τεχνικών εμπειρογνωμόνων, ε, μελών πολιτικής ή ε, συμβούλων κυβερνητικών που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, με συγκεκριμένες και χρήσιμες συμβουλές. Θέλουμε να καταρτήσουμε και το στρατιωτικό και το πολιτικό σκέλος, για τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν, ε, για την αλληλοκατανόηση και την κατανόηση των συστημάτων τους. Θέλουμε να βοηθήσουμε κάθε κράτος να αντιμετωπίσει μια κυβερνοεπίθεση και να λάβει σωστές αποφάσεις και από διπλωματική και από νομική άποψη. Στόχος μας είναι να ασκήσουμε πίεση στις ομάδες στα επιτελεία και να τα δοκιμάσουμε σε όρους μιας μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης, απευχόμενη φυσικά την ε, πραγματικότητα αυτή. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε τις ομάδες αυτές για να ανταποκρίνονται στις τεχνικές εξελίξεις ε, με ε, εύληπτο τρόπο. Επίσης, παρέχουμε μελέτες για το τι συμβαίνει προκειμένου να στέλνονται από τους εμπειρογνώμονες στις κυβερνήσεις και έχουμε γίνει επανειλημμένοι μάρτυρες αυτού του τροτού σημείου της κυβερνοασφάλειας, της κοινότητας κυβερνοασφάλειας. Επίσης, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια νομικά ζητήματα, γιατί το νομικό πλαίσιο του, της δικτυοπαραβίασης και του υβριδικού πολέμου είναι ασαφές. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η κλίμακα και τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ε, όταν απλώς ε, καταρρύπτεται, ε, χρηστεύεται μια σελίδα επιχείρησης, δεν θεωρείται υβριδικός πόλεμος, αλλά αν παραβιαστεί η μια βάση πυράβλων είναι αλλιώς τα πράγματα. Επίσης, ανταπόκριση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο σκέλος που αφορά τα ΜΜΕ. Θα πρέπει να μπορούν τα μέλη μας, δηλαδή μάλλον τα μέλη αυτών των ομάδων, να παρουσιάζουν ε, το θέμα στα μίδια με σωστό τρόπο. Τώρα, ποια είναι η αξία αυτών των ασκήσεων, αυτών των γυμνασίων. Θεωρούμε ότι τέτοια ασκήσει μεγάλη κλιμακό, όπω είναι το Cyber Coalition ή το Locked Shields, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία για τις εθνικές ομάδες ε, να συμμετέχουν και να παρακολουθούν πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε τέτοιου είδους ε, κυβερνοσύγκρουσης. Και πραγματικά αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Ποια είναι τώρα η συνταγή της επιτυχίας. Πρώτα απ' όλα το κλειδί είναι να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες και να έχουμε πάντα μια γενική εικόνα της κατάστασης. Επίσης να προσαρμόσουμε την αρχική αμυντική στρατηγική στις εξελίξεις. Για παράδειγμα, ε, τα σενάρια που εξετάζουμε στο Lock Shields ε, μας προετοιμάζουν για τις μελλοντικές επιθέσεις, χάρη στην κατάρτιση που προσφέρουμε. Επίσης, η Εστονία που μας φιλοξενεί έχει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κυβερνοάμυνας και από πρώτο χέρι μάλιστα. Γιατί υπέστη μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων το 2007 που έδωσε λαβή για την πρώτη σοβαρή και εκτεταμένη δημόσια συζήτηση για το πιθανό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν κυβερνοεπιθέσεις στην εθνική ασφάλεια τα μαθήματα που αντλήσαμε από τις επιθέσεις αυτές ήταν ότι η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων εντοτήτων, όχι μόνο στρατιωτικών, αλλά και κυβερνητικών και πολιτικών, αλλά και μεμονωμένων πολιτών. Ένα έθνος κράτος ε, φυσικά είναι κυρίως αρμόδιο για την ανέβρεση λύσεων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν κάποιο ρόλο και μπορούν να προσφέρουν αρρωγή. Τα γεγονότα του 2007 επιλήθηκαν χάρη στη συνεργασία. Ένας συλλογικός εγκέφαλος ε, από, με δημόσιες και ιδιωτικές πτυχές ε, συνεργάζονταν με σύμπνια. Θεωρούμε ότι οι ασκήσεις επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ενημερωθούν για τις ε, δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που έχουν. Και μια πανευρωπαϊκή άσκηση δεν είναι μια, κάτι το ανέφικτο, αλλά μια επιτακτική ανάγκη για να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μόγκρε. Και τώρα, σύμφωνα με τους κανόνες μας, προτείνω στις ομάδες, στους κοιόδης εισηγητές, να λάβουν το λόγο για δύο λεπτά ο καθένας. Μετά, άλλα ενδιαφερόμενα μέλη θα μπορούσαν να μιλήσουν για ένα λεπτό και μετά οι θα απαντήσουν στις σα ερωτήσει. Και οι δύο θα έχουν πέντε λεπτά. Οργανισμός ΕΝΗΣΑ, ο κ. Πέρσερ, επικεφαλής στο τμήμα της συνεργασία. δύο λεπτά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Δέσπινα Σπανού για τρία λεπτά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμά μας. Η κυρία Αγγέλικα Νίμπλερ, ο πλευρά ΣΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που διέθεσαν το χρόνο τους και μας ωφέλησαν μέσω μετάδοσης της τεχνογνωσίας τους και της εμπειρίας τους. Θα είμαι τάχιστη. Πολύ καλή γενική εισαγωγή αυτή που ακούσαμε για το θέμα. Σαφώς η Ευρώπη μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά την κυβερνά ασφάλεια. Και σαν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου εμεί πρέπει να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι κρίσιμες ε, κριτικές υποδομές, οι κρίσιμες υποδομές όπως είναι το διαδίκτυο, θα λειτουργούν σωστά και θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια για τους απλούς πολίτες, για τους κυβερνητικούς φορείς και για τις επιχειρήσεις. Ασφάλεια στο διαδίκτυο και πιστεύω ότι η υποβληθήσα πρόταση είναι πολύ καλή, πολύ λογική. Η ΕΝΗΣΑ χρειάζεται περισσότερους πόρους, ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους. Και είναι σημαντικό να δοθεί μια σαφέστατη εντολή στον οργανισμό αυτό και να τύχει της δέουσας υποστήριξης και να έχει την κατάλληλη θέση που της αρμόζει. Τώρα πηγαίνουμε στον τομέα της πιστοποίησης. Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που γίνονται για την πιστοποίηση εγώ δεν έχω κάποια ξεκάθαρη ιδέα όσον αφορά το θέμα αυτό και πώς θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών μέλων και Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά είναι καλή ευκαιρία αυτή να διερευνήσουμε το θέμα αυτό. Ακούσαμε σήμερα ποια είναι η κατάσταση. Μας το εξήγησε ο κύριος Σάπχουσα δεν είναι κάτι που αφορά όμω μόνο τη Γερμανία, υπάρχουν και άλλα 27 κράτη-μέλη εκτό Γερμανία. Ερώτηση. Βλέποντα ε, τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα, ποια είναι η άποψή σα. Θεωρείτε ότι οποιοδήποτε ρόλος ανατίθεται στην ενίσα θα οδηγήσει σε πίεση όσον αφορά τους ε, υπάρχοντες ε, οργανισμούς σε ένα δικτυωμένο κόσμο. Η Γερμανία ενδεχομένως να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά το θέμα. Πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται και με την ασφάλεια των άλλων 27 χωρών. Και ίσως υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων που έχουν οι άλλες χώρες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει την εσωτερική αγορά, πρέπει να είναι βέβαιος ότι το επίπεδο κυβερνασφάλειας είναι πολύ υψηλό. Και αυτό ισχύει και για την πιστοποίηση, διότι η κυβέρνοασφάλεια μπορεί να είναι δύσκολο θέμα να επιληθεί, αλλά μας δίνει ε, καλή θέση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ο Πέτερ Κρούμπασεφ, ε, που είναι σχεδόν συγγητής για τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, αυτά που είπε ο κύριος Σέφερ, κυρίως στο τέλος, που είπε ότι ίσως δεν θα πρέπει να βάζουμε πολλές ελπίδες στον οργανισμό τον ευρωπαϊκό της Κυβερνασφάλειας, είπε ο κύριος Απρούζερ. Για να έχουμε έναν ισχυρό φορέα για την κυβερνασφάλεια στην Ευρώπη, θα πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ε, τα εθνικά όρια και τους εθνικούς εγωισμούς, την εσωστρέφεια των διαφόρων υπηρεσιών, που ε, προβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, κύριε Σάπχουζα, πιστεύετε ότι οι εθνικοί οργανισμοί και υπηρεσίε θα πρέπει να διατηρήσουν τι αρμοδιότητε που έχουν. Και ποιε αρμοδιότητε θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να τεθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Για να έχουμε έναν αποτελεσματικό οργανισμό, πρέπει ο οργανισμό να έχει σοβαρότατε αρμοδιότητε. Και όχι να είναι ένα εικονικό ιονή οργανισμό που εμφανίζεται ότι είναι υπεύθυνο για την κυβερνοασφάλεια, αλλά ουσιαστικά έχει απλώς ενημερωτικό ρόλο. Δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών, οργανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς να έχει πραγματικές δυνατότητες και εξουσίες να δράσει. Τώρα μια ερώτηση προς την κυρία Μέγκρε. Σας ευχαριστώ καταρχάς που παρουσιάσατε τα όσα κάνει το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ καλό το ότι γίνονται συγκεκριμένα πράγματα. Η ερώτησή μου αφορά το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων. Θεωρείτε ότι η δική σας διεύθυνση, το τμήμα σας, το κέντρο σας μάλλον, στην Ενίσα, και η Ενίσα μπορούν να συνεργαστούν. Διότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και στον τομέα της συνεργασίας. Υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν εγωιστικές τάσεις σε επίπεδο κρατών μελών, διότι υπάρχουν διάφοροι φορείς στα διάφορα κράτη που δουλεύουν διαφορετικά και όλα αυτά οδηγούν σε επικοινωνία που δεν είναι η αρμόζουσα και η επιθυμητή. Δεν έχουμε κοινή δράση. Εμείς θα θέλαμε κοινή δράση στο μέλλον. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρίτος, για το ECR, ο κ. Σινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη διοργάνωση της ακροάσεως αυτής για την ασφάλεια. Διότι με την επέκταση της πληροφορικής και των συναφών συστημάτων, ο αντίκτυπος προβλημάτων στα, στις υποδόμες ε, πολλαπλασιάζεται. Έχουμε περίπλοκα συστήματα και επειδή είναι περίπλοκα τα συστήματα, ε, είναι επιρρεπή τα συστήματα σε επιθέσεις. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεγιστοποιήσουμε την αντίσταση αυτών των συστημάτων στις επιθέσεις. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Την επιθύνω στον κύριο Σαπχούζερ. Και εγώ πιστεύω ότι η ΕΝΙΖΑ πρέπει να ενισχυθεί. Όμως θα προτιμούσα η ΕΝΙΖΑ να παίζει περισσότερο το ρόλο συντονιστού, ένας συντονιστής υψηλού επίπεδου, διότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν μεγάλο οργανισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω να διαθέτει εμπειρογνώμονε που μπορούν να καλύψουν κάθε πτυχή του προβλήματο. Ένας τέτοιο οργανισμό πολύ γρήγορα θα έχανε έδαφο διότι θα κατέρε, θα, θα είχαμε εσόριξη του οργανισμού λόγω του μεγάλου του βάρους. Θα πρέπει νομίζω να χρησιμοποιήσουμε τους εθνικούς φορείς και να ενισχύσουμε τα δίκτυα εμπειρογνωμόνων και τους ιδιωτικούς ε, ανάλογους φορείς. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε εθνικό επίπεδο πάντα. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργούσε ένα τέτοιο μοντέλο και πώς βλέπετε το βαθμό συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, διότι αυτού του είδους οι υπηρεσίες συνήθως δεν θέλουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Δεν τους αρέσει πολύ αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. δεύτερη ερώτηση. Η συνεργασία μεταξύ των υφισταμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πώς πάει το Κοινό Κέντρο ερευνή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η Ευρωπόλ, ε, πώς συνεργάζονται, διότι έχουν και αυτοί οι φορείς πολλές αρμοδιότητες στον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Αντί την κυρία Ταρίσκα ε, Λοιπόν, Thank you for the introduction. ακούσουμε την κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγκράτησα από αυτά που είπε ο κύριος Σαμπχούζα στην παρουσίασή του ότι τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητες και θα έπρεπε να τις έχουν, διότι τα συστήματα πληροφορικής τα χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Οπότε εκεί θα πρέπει να παραμείνει η αρμοδιότητα, στα κράτη-μέλη. Η κυρία Μέρνε Μάγκρε αναφέρθηκε στο θέμα της γενικής εικόνας. Πώς μπορούν να καταπολεμηθούν τα προβλήματα με μια κοινή προσπάθεια. Έχω μια ερώτηση. Αν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ των φορέων, εάν θα πρέπει να γίνονται περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ενίσα, σε σχέση με τους εθνικούς φορείς. Πώς σχηματίζουμε τη γενική εικόνα αν πολεμάει κάθε χώρα ξεχωριστά το πρόβλημα. Τα κάτι μελη έχουν πρόβλημα στο να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι οι κακοί μοιράζονται τις πληροφορίες, ενώ οι καλοί δεν τις μοιράζονται. Αν κάποιος δεχτεί κυβερνοεπίθεση, κάποιος άλλος θα μπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες και να μάθει αν πληροφορηθεί. ή αν συνεργάζονται και εταιρείε και ενημερώσει μια εταιρεία την άλλη ότι έχει υποστεί επίθεση και άλλη έτσι να προστατευτεί. Ερώτηση. Αν είμαστε αντίθετοι στην ευρωπαϊκή προσέγγιση, να δράσει ο οργανισμό εν ίσα, πώ θα κάνουμε, θα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, τόσο ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ε, greens. Από τους πρασίνους παρακαλώ κανένας δεν βρίσκεται στην αίθουσα παρόν, από το ΙΕΝΕΦ, e Κρίστε Λεβασουριέ, ή κάπως έτσι. Η Λεσεβαλία διορθώνει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, δεν ζήτησα το λόγο. Ακούω και παρατηρώ. Καλώς. Οπότε Θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Η κυρία Καηλή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας που σχολίασαν ε, την έντολη του ΕΝΙΣΑ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο και βασικό βήμα για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις κυβερνοαπειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μιλήσατε και για την πιστοποίηση, για να αυξήσουμε την κυβερνοασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έχω κάποιες απορίες. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση σημαντικής κυβερνοεπίθεσης, μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, τι δυνατότητες έχει ο ΕΝΙΣΑ να διεκπαιρεώσει το έργο του και το επιχειρησιακό του ρόλο χωρίς παρέμβαση των κρατών μελών ώστε όχι να συντονίζει απλώς, αλλά να αναλάβει επιχειρησιακό ρόλο πολύ πιο συγκεκριμένο σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Επίσης, τι γίνεται με τις ε, κυβερνοδεξιότητες, ε, Ήδη στο σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να δίνονται πληροφορίε και γνώσει για το πώ μπορούμε να προστατευτούμε από κυβερνοεπιθέσει. Οπότε έχουμε πολλέ προκλήσει που αφορούν και τι νέε τεχνολογίε. Δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα των δεδομένων και την κυβερνοάμυνα, αλλά περνάει σε θέματα τεχνητή, νοημοσύνης, ρομποτική και ούτω καθεξής. Πιστεύετε ότι και αυτά θα περιληφθούν στο διευρυμένο ρόλο του ΕΝΙΣΑ, γιατί είναι πολύ άριθμες οι προκλήσεις. Και αν αυτό παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών και από τη στιγμή που το διαδίκτυο δεν γνωρίζει σύνορα και οι απειλές είναι οικουμενικές και οι αντιδράσεις μας αυτές τις απειλές θα πρέπει να είναι καθολικές. Πώς βλέπετε επίσης τη συνεργασία του ΕΝΙΣΑ με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Καϊλή. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μούντι. Όχι, δεν θέλει, δεν τον ζήτησε. λαμπρά. Ο κύριος Ζωχρίνιο, ούτε και αυτός. Τέλεια. Οπότε ήδη ακούσαμε τις ερωτήσεις όλες. Τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, τον κύριο Σαπχόιζερ και την κυρία Μόγκρε, για να απαντήσει στην πληθώρα των ερωτήσεων των συναδέλφων. Να προσθέσω και εγώ τη... κάτι. Ε, δεν έχουμε μόνο την κατάσταση στο συγκεκριμένο αυτό κλάδο. Το έχουμε και στο θέμα του ηλεκτρισμού και σε άλλες υπηρεσίες. Γιατί η προστασία των δεδομένων είναι ένα είδος παροχής υπηρεσίας. Και είναι σημαντική ευθύνη των κρατών εθνών και για τους πολίτες. Πώς όμως θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός από τον ΕΝΙΣΑ, ο καλύτερος συντονισμός αυτών των δραστηριοτήτων καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε δεξιότητες και να προβλέψουμε κατάρτιση για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απειλές. Μας είπατε το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει εμπειρογνώμονες για τέτοια θέματα. Αλλά άλλο το στρατιωτικό σκέλος του προβλήματος και άλλο το πολιτικό. Γιατί οι περισσότεροι πολίτες επιθυμούν γενικώ προστασία των δεδομένων. Έχουμε όμως παροχή ενέργειας, μεταφορές και εκεί τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και ευάλωτα στην κυβερνοαπειλή. Παρακαλώ, κύριο Σάπιουιζερ. Ο κύριο Σάπιουιζερ, θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, ε, στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, ε, μάλλον δήλωση, εμείς του BSE, του γερμανικού BSE, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του ΕΝΙΣΑ η εκτίμηση για το ποια είναι η θέση των υπολείπων χωρών μελών της Ευρώπης ό,τι αφορά τη δημιουργία πρόσθετων δομών, θεωρώ ότι χρειάζεται πράγματι μια ανάπτυξη του τομέα αυτού σε πολλές χώρες μέλη. Όμως θεωρώ ότι είναι κατεξοχήν αποστολές που είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Εκεί ο ρόλος του ΕΝΙΣΑ μπορεί να είναι παροχή συμβουλών, παροχή κατευθύνσεων. Θα έρθω πάλι στο θέμα αυτό Για την ερώτηση σχετικά με τους ισχυρούς εγωισμούς των χωρών μελών. Εγώ δεν βλέπω τον Ενίσα ως ανταγωνιστή. Βλέπω τον ρόλο του υποστηρικτικό για την εξασφάλιση ε, για την εγγύηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στη Γερμανία. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, για παράδειγμα, εποπτεύονται από εθνικούς οργανισμούς. Οποιαδήποτε κρίση κυβερνοασφάλειας αναφέρεται αμέσως στις εθνικές αρχές. Επομένως είναι πάρα πολύ ισχυρός αλλά και αναγκαίος ο ρόλος των ε, χωρών μελών στην αντιμετώπιση των κρίσεων ασφάλειας. Για τον καλύτερο συντονισμό, ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν υπάρχει ψηφιακός κόσμος και αναλογικός κόσμος. Υπάρχει ένας ενίος κόσμος και ο κόσμος αυτός είναι όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένος. Επομένως δεν μπορούν να διακρίνονται οι διαδικασίες προστασίας της ασφάλειας. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ΕΝΙΣΑ. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό μάλιστα, πολύ σημαντικός ο ρόλος της παροχής πληροφοριών. Capacity building, διεξαγωγή ασκήσεων. Συμφωνώ με την συνάδελφό μου κυρία Μόιγκρε ότι είναι από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη για να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε κρίση. Γιατί μόνο μέσω των ασκήσεων βρίσκει, εντοπίζει κανείς τα αδύναμα σημεία του συστήματος. Το ερώτημα της συνεργασίας μεταξύ των διαφορών αρχών και μνημονεύτηκε εδώ η Ευρωπόλ. Εγώ θεωρώ ότι ο τομέας του κυβερνοεγκλήματος αντιμετωπίζεται από το Εθνικό Ποινικό Δίκαιο και παραπέμπεται στην Ευρωπόλ. Δεν θεωρώ ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να στραφούν πρώτα στον Ενίσα και μετά στην Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ στην βάση πληροφοριών που θα διαθέτει μπορεί να παραπέμψει παραπέρα στον ΕΝΙΣΑ και στην ε, Cyber Security Community γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το γενικότερο σύνολο, κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά μετριοπαθή σχετικά γιατί 26 χρόνια έχω ε, ασχοληθεί με θέματα κυβερνοασφάλειας και έχω μάθει να είμαι πάρα πολύ μετριόφρον. Προέτους εκδόθηκε η οδηγία NIS. Σημαντικό είναι να εφαρμοστεί σοβαρά και να προβλέπει μέσα και capacity building και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να ενισχυθεί το disaster recovery, χρειάζεται να ενισχυθούν οι δομές αντιμετώπισης, βεβαίως χρειάζονται πολύ σημαντικό συντονισμό και εκεί ο ΕΝΙΣΑ μπορεί να παίξει ένα πολύ κεντρικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τώρα την πιστοποίηση, θεωρώ επίσης ότι Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πιστοποίησης. Ωστόσο, οι υφιστάμενες δομές να εξελιχθούν προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς να γίνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο εμπόδιο στις προσπάθειές τους. Ο ΕΝΙΣΑ τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί με ρομποτική, αλγοριθμική και ούτω καθεξής. Τι να σας πω, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Εμείς το μελετούμε ακόμα, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσουμε είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να είναι μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια, γιατί η ισχύ των αλγορίθμων θίγει όλους. Μπράβο, σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τον ε, χρόνο των πέντε λεπτών που σας διέθεσα. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στις κρίσιμες υποδομές σε μια ερώτηση. Όντως, οι κρίσιμες υποδομές έχουν κομβικό ρόλο στην οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια των κρατών μας και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ένα στρατιωτικό και ένα πολιτικό σκέλος στην ασφάλεια, με τις εθνικές υποδομές φυσικά να είναι στο στόχαστρο των κυβερνοεπιθέσεων. Τι μας ανησυχεί, τα, τα δίκτυα ενέργειας, ε, πλοήγηση, τηλεπικοινωνίες, ε, νοσοκομεία, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταφορές. Όλα αυτά τα συστήματα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και θα ήταν ίσως βολικό να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ της στρατιωτικής διάστασης και των κρίσιμων εθνικών υποδομών δεν είναι εύκολη μια τέτοια διαχωριστική γραμμή, γιατί χρειαζόμαστε αναφυσβήτητα στρατιωτική και μη στρατιωτική συνεργασία. Γι' αυτό σας είπα δεν πρέπει να χαθούμε σε λεπτομέρειες και να δημιουργήσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Ε, και αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο σκέλη και κυρίως χάρη σε αυτές τις πρακτικές ασκήσεις που οργανώνουμε. Τις ασκήσεις ε, που οργανώνονται ε, και προϋποθέτουν τη συνεργασία των κρατών μελών και τη συμμετοχή τους ε, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Και εκεί συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και μετά αξιοποιούν ή την έκθεση ή τα συμπεράσματα που αντιλήσαμε από τις ασκήσεις και τα εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που προέχει εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε σενάρια ε, που περιγράφουν την πραγματικότητα, ώστε να μην νιώθουν τα κράτη ότι είναι αφηρημένες αυτές οι ασκήσεις ε, και αφηρημένες οι προσωμιώσεις. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούν επιχειρησιακά συστήματα που θα συναντήσουν και στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα. Μόνο έτσι θα δοκιμάσουμε τις πραγματικές ουσιαστικές δεξιότητες και θα δημιουργήσουμε ουσιαστικές ικανότητες για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απειλές. Οπότε δύο θα ήταν τα συμπεράσματά μου. Δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει θαυματουργή λύση, αλλά υπάρχει ανάγκη χαρτογράφησης και σύγκρισης και τον μηχανισμό διαχείρισης, διαχείρισης κρίσεων της κυβερνοασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να βρούμε δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας. Έτσι θα, θα ενισχύσουμε την κοινή ε, αντίληψη της κατάστασης σε θέματα κυβερνοασφάλειας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός, γιατί πολλά ήδη έχουν γίνει και προηγηθεί, οπότε θα πρέπει να στηριχθούμε στη χαρτογράφηση και στις ε, εμπειρίες μας από τις ε, ασκήσεις που κάναμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το EU Cybrid για παράδειγμα, που έγινε για πρώτη φορά σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας φέτος, το Σεπτέμβριο, τις παράλληλες και συντονισμένες ασκήσεις της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκήσεις του ΝΑΤΟ για διαχείριση των κρίσεων που φέτος επικεντρώνονται στις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και το Cyber Europe που οργάνωσε ο ΕΝΙΣΑ και οργανώνει κάθε διετία. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια χαρτογράφηση της συνεργασίας μας με βάση τις ανάγκες κυβερνοασφάλειας και με βάση τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από τις μέχρι τώρα ασκήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει για να βελτιώσουμε τη συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, θα πρέπει να εντοπίσουμε ε, τις ανάγκες κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας ε, που είναι χρήσιμες και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την 1η Πρώτου 2018 το Κέντρο Αριστείας μας θα αναλάβει ε, το ρόλο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΝΑΤΟ για την κυβερνοασφάλεια για να αναλύσουμε τις ανάγκες που έχει η Συμμαχία για την κατάρτιση σε τέτοια θέματα και να ανταλλάξουμε και να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μόνη ερώτηση που δεν απαντήθηκε μέχρι τώρα, δηλαδή τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ίσως θα μπορούσε να απαντηθεί από τον Steve Purser επικεφαλής του Τμήματος Συνεργασίας. Έχετε το λόγο λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εν είδη αγωγής, να πω ότι πολύ ευπρόσδεκτη δέσμη μέτρων, πολύ φιλόδοξο πακέτο και ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Είναι απαραίτητο κατά την άποψή μας παρακολουθείτε τις διάφορες στοιχές του προβλήματος και θα συμφωνείτε ότι πρέπει τα βήματα που θα κάνουμε τώρα να είναι φιλόδοξα και κάνουμε τώρα ευπρόσδεκτο το πακέτο και η εντολή και οι πόροι που είναι απαραίτητοι για μας ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε σταθερότητα, να εκμεταλλευτούμε τα επιτευθέντα όσον αφορά τις υποδομές πληροφοριών και ενημέρωσης και να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τα νέα προβλήματα. Το ερώτημα αφορούσε τη συνεργασία. Να υπενθυμίσω κάτι. Υπάρχει σημαντικό επίπεδο συνεργασία. Εγώ είμαι στο Συμβούλιο το Αρμόδιο, ε, το οποίο συντονίζει τις δραστηριότητες στον τομέα. Μοιραζόμαστε πληροφορίες με δυναμικό τρόπο. Και τώρα, και κάτι άλλο που συμβαίνει κάθε χρόνο, έχουμε την ε, μεικτή συνεδρίαση της ΕΝΙΣΑ, Europol, EC3 και ε, μοιραζόμαστε πληροφορίες εκ μέρους των διαφόρων φορέων. Μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Καλή ιδέα που ακούστηκε να υπάρχει διαβίβαση πληροφοριών και συνεργασία με το CCCDE και συμμερίζομαι και αυτή την άποψη περιασκήσεων. Ε, είναι πολύ καλός τρόπος οικοδομήσεως εμπειρίας και χρήσεως της εμπειρίας για βελτίωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και για την εφαρμογή μελλοντικών λογικών πολιτικών. Αυτά είναι τα κρίσιμα σημεία και κάτι άλλο. Η Ενίσα πάντα ήταν και θα είναι ένας οργανισμός που αφορά τη συνεργασία. Ό,τι κάνουμε αφορούν την καταλητική μας ιδιότητα να βοηθούμε τους φορείς να συνεργαστούν. Εμείς έχουμε στόχους για την ευρύτερη κοινότητα, όχι μόνο για τον οργανισμό μας. Και το λέω σοβαρά. Άρα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ε, κλίμακα, έχουμε 50 άτομα προσωπικό που είναι άριστο προσωπικό, δεν αλλάξουμε τον κόσμο όμω. Όταν όμω μοιραστεί την τεχνογνωσία σου με το κάτι μέλη, τότε έχει παραπλασιατικό αποτέλεσμα. Αλλάζει κλίμακα. Και ε, προσετερίζονται, χρησιμοποιούν αυτά τα αποτελέσματα τα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και κινούμεθα προ το τελικό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό το μήνυμα για το μέλλον. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση στο μέλλον. Θέλουμε πολύ περισσότερη συνεργασία. Προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία και ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος. Μία απλή ερώτηση που δεν απαντήθηκε όμως. Βαθμός συνεργασίας μεταξύ 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης δεν σπινάς πανού που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια ε, να απαντήσει για αυτό το θέμα το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Έχουν υποβληθεί προτάσει. Εμεί θέλουμε να βοηθήσουμε του συνομοθέτε και να προβούμε στι διευκρινήσει. Στα όσα υπόθηκαν και όσον αφορά και την ερώτησή σα. Η προτινόμενη εντολή βασίστηκε σε απλούστατη βάση. Καταρχά, το έργο τη ΕΝΗΣΑ. Δημιουργία δυναμικού, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, διαβίβαση των των ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, όπως είπαν και διάφοροι προλαλήσαντες ομιλητές. Και μετά να βασιστούμε και σε στήματα δικτύωσης και πληροφορικής και τη σχετική οδηγία και τον, την νομοθεσία περί ασφαλεία. Σημαντικό όταν εξετάζουμε το θέμα της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ επίπεδου κρατών μελών και του οργανισμού, διότι δημιουργήθηκε καταρχάς ένα δίκτυο ομάδων, το ΣΥΣΕΝ δίκτυο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και εκεί αναφέρεται η ενίσχυση ότι έχει σημαντικό ρόλο να παίξει εκεί, διότι είναι η γραμματεία του δικτύου αυτού για την ασφάλεια. Ήδη από την προηγούμενη θητεία, την προηγούμενη νομοθεσία, προβλέπεται ενίσχυση τη ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή και τη αντοχή τη και να βοηθηθεί η γραμματεία και το δίκτυο των κρατών μελών που κάνει τη δουλειά του. Ήδη υπάρχει καλό συντονισμό λοιπόν μεταξύ κρατών μελών. Τι κάνει η πρόταση. Κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, καθορίζει λεπτομερώς τα καθήκοντα του οργανισμού. Είναι μικρός οργανισμός σε κλίμακα, με συγκεκριμένο ρόλο και μπορεί να πετύχει τους στόχους του και να εκτάσει τα καθήκοντά του θέλουμε, αυτό θέλουμε. Και έχουμε επιχειρησιακή ε, συνεργασία του SIS Network και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην ε, ΕΝΗΣΑ να βελτιώσει τη δυνατότητα ανταπόκριση των κράτων μελών, κατόπιν αιτήματος αυτών θα παρέχεται η τεχνική αρρωγή σε περίπτωση επεισοδίων. Δεν αντικαθιστά η τι ομάδε ανταπόκριση των κρατών μελών, αλλά βοηθά μέσω τη τεχνογνωσία τα κράτη-μέλη που ίσω χρειαστούν κάποια βοήθεια και τη ζητήσουν τη βοήθεια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή που έχει σημαντικό ουσιαστικό αντίκτυπο. Να αναλυθούν οι ευαισθησίε, τα διάφορα επεισόδια. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα για να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση και η Ευρώπη περί αντιμετωπίσεω προβλημάτων κυβερνοασφαλείας. Επουδενή δεν είναι μια πρόταση που απαιτεί αντικατάσταση των εντολών των εθνικών φορέων για την κυβερνοασφάλεια. Αντιθέτω, μάλιστα, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε όταν αυτό χρειαστεί και απαιτηθεί και αν είναι αναγκαίο του εθνικού φορεί και θα είναι κόμβο συγκέντρωση δημιουργία τεχνογνωσία και δυναμικού για όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα ερχόμενοι στις πιστοποίησεις. Γιατί προτείναμε την ενίσα στον κανονισμό. Διότι είναι ένα τυπικό καθήκον ενός ανεξαρτήτου ευρωπαϊκού οργανισμού σε αυτό το μόρφωμα που προβλέπουμε. Έχουμε έναν ανεξάρτητο φορέα που έχει τεχνογνωσία. Η ενίσα ήδη έχει εργαστεί επί πιστοποίησεων και στην πιστοποίηση της νεφοϋπολογιστικής cloud Οπότε βασίζεται στην υφιστάμενη τεχνογνωσία, αλλά αυτό δεν αφαιρεί το ρόλο των κρατών μελών. Να σας εξηγώ τι προτείναμε. Είναι, κάνει εξολόγηση προτάσεων ευρωπαϊκών σχημάτων η ΕΝΗΣΑ, τα προτείνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά είτε τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους και τα κράτη-μέλη ψηφίζουν για την έγκριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πιστοποίησης ε, με τη δικασία των εφαρμοστικών πράξεων και τέλος κατεξίσου σημαντικό τώρα στον συνεργασία. Πράγματι σε αυτή την πρόταση καθορίζουμε τη δομημένη συνεργασία που θα πρέπει να έχει ενίσα με τους άλλους φορείς, να αποφύγουμε επικαλύψεις του το τρόπος και στο σχέδιο που προτείνουμε και τις συστάσεις του στα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση επεισοδίων μεγάλης κλίμακας καθορίζουμε και το ρόλο του κάθε φορέα επακριβώς, ούτως ώστε το σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικός πως. Αυτό το σχέδιο θα δοκιμαστεί στην άσκηση που θα γίνει το 2018 ε, αναφέρθηκε ήδη αυτή η άσκηση ότι είναι κάτι σημαντικό για να τροφοδοτεί η τεχνογνωσία τη ΕΝΗΣΑ και προτείναμε ότι αντί αυτό να γίνεται κάθε δύο χρόνια, αυτή η άσκηση να γίνεται ετησίω. Λυπάμαι που ξεπέρασα τα χρονικά μου όρια, αλλά ελπίζω να απάντησα στι ερωτήσει. Καλώ. Ευχαριστούμε. Περάσετε με τα σχόλιά σας ε, και στο δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασης. Κάνατε μια πολύ καλή μετάβαση, γιατί σε μερικές απαντήσεις καλύψετε ζητήματα του δεύτερου τμήματος της ακρόασης. Θα σας ε, παρουσιάσω τους καλεσμένους μας για το δεύτερο τμήμα. Θέμα είναι η κυβερνοασφάλεια και το σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος μας ομιλητής για το τμήμα αυτό είναι ο κύριο Γκαμπριέλε Φατζόλη, ε, πρόεδρος της Κλούσιτ ε, του Ιταλικού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Υπολογιστών ε, καταρχήν το υπόβαθρο, το επαγγελματικό πρόεδρο ε, του οργανισμού Κλούση, του Ιταλικού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Υπολογισμών. Επίση είναι επιστημονικό διευθυντή ε, στο, στη Σχολή Διοίκηση του Πολυτεχνείου του Μιλάνου με θέματα ασφάλεια και πληροφορία, ιδιωτικές πληροφορίες. Είναι διευθυντής του Partners for Innovation, μιας επιχείρησης που είναι υποκατάστημα του Digital 360 που είναι καταχωρημένη και στο τελικό χρηματιστήριο και είναι εταίρος και ε, φορέας διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Φαντζόλη είναι εμπειρογνώμων και ειδικό για νομικές πτυχές της ασφάλειας των υπολογισμών. Οπότε έχετε το λόγο για το σύστημα πιστοποίησης της, για την κυβέρνηση ασφάλεια. Θα περιμένουμε τις φαϊνές σας προτάσεις και ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε όλοι. Είμαι ο Γκαμπριέλε Φατζόλη και είμαι ο πρόεδρο τη Κλούζη τη Εθνική Ένωση για την Ασφάλεια των Υπολογιστών. Η Κλούζη είναι ο σημαντικότερο οργανισμό τη Ιταλία. Θέλουμε να υπερασπιστούμε και προωθήσουμε ε, την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων, των εταιριών, των πολιτών και τη δημοσιοδιοίκηση Και επίση είμαι επιστημονικό διευθυντή ε, του παρατηρητηρίου τη ασφαλεία του Πολυτεχνείου του Μιλάνου και διαδίδουμε τεχνογνωσίε για δυνατότητε ε, και προκλήσει που έχουμε από πλευρά τη ε, ψηφιακή τεχνολογία για τι επιχειρήσει, τη δημόσια διοίκηση και για του πολίτε. Πριν αναλύσω ε, λεπτομερώ τι διάφορε διατάξει του νέου κανονισμού, θα ήθελα να πω ότι το, αυτό το σχήμα τη πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση ανταγωνιστικότητα και τη καινοτομία και να έχουμε ασφαλέστερο χώρο. Η αξία του προγράμματο πιστοποίηση αξίζεται σε δύο βασικού όρου. Καταρχά, θα πρέπει εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά να υθετήσουν αυτά τα σχήματα και δεύτερον θα πρέπει οι χρήστες να αναγνωρίσουν την αξία που έχει. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σχήμα πιστοποίησης να έχει σαν ένα στόχο που να μπορούν να, να επιτευχθεί. Λοιπόν, θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο κυβερνοασφαλείας σε υψηλότερα επίπεδα. Οι καλές πρακτικές και η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζουν στόχου ε, βάσει μειώσεω του κινδύνου και όχι απλώ επίπεδο ε, εξασφάλιση από τον κίνδυνο. Η κυβερνοφάρεια σήμερα είναι ένα από του παράγοντε που προτιμά, προστατεύει την αξία, τα συμφέροντα των πολιτών όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίε. Θα πρέπει να προσέξουμε αυτή την πτυχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τότε τα αγαθά και υπηρεσίε τελικά θα είναι πιο ελκυστικά κυρίω ε, για τι νέε αγορέ και, ε, και αγορέ ψηλή αξία. Θέλουμε να βελτιώσουμε και για τι εταιρείε και για του πολίτε την κυβερνοασφάλεια. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σύστημα πιστοποίηση που ασχολείται με αυτού του κινδύνου ε, θα μπορούσε να βοηθήσει. Η κυβερνοασφάλεια αλλάζει καθημερινά μαζί με τι νέε τεχνολογίε και τι νέε επιθέσει. Άρα χρειάζεται μια μεγάλη έρευνα και περισσότερε επενδύσει όσον αφορά την καινοτομία. Η σημερινή πρόταση για κάποιον κανονισμό καθορίζει μια σειρά διαφορών στοιχείων για την αποφυγή και πρόληψη ενδεχόμενου κατακαιρματισμού των συστημάτων πιστοποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτέ τι προτάσει έχουμε ένα νοητικό πλαίσιο για κανόνε που διέπουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα τη Πιστοποίηση και και είναι ένα πλαίσιο που θα πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένα συστήματα πιστοποιήσεω για διάφορα προϊόντα ασφαλεία, που πρέπει να καθορίζονται οι συνθήκε και όροι. Ξέρουμε ότι η πιστοποίηση είναι η επίσημη αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και διαδικασιών που θα πρέπει να τα σέβεται κάθε φορέα όσον αφορά διάφορα κριτήρια σταθερά. Και για αυτού του λόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινηθούμε στον τομέα των ε, υπολογιστών. Για την ασφάλεια υπολογιστών στον τομέα. Επί παρόντο, η Ευρωπαϊκή Θέση την κυβερνοασφάλεια και την πιστοποίηση για τα προϊόντα τη πληροφορική είναι κατακαιρματισμένη η κατάσταση οδηγεί σε αύξηση του κόστους και είναι οικονομικό άχθος για εταιρείε που λειτουργούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Τελικό στόχο, ε, απότοτο στόχο τη προτάσεω είναι να προσφέρει ωφέλη στου πολίτε και στι επιχειρήσει. Ε, σύμφωνα με την άποψή μου, θα πρέπει να θετηθεί μια διαφορετική προσέγγιση που θα εδράζεται επιμειώσει του κινδύνου στην πρόταση, σύμφωνα με τι τεχνικά πρότυπα βιομηχανία ISO 27001, παραδείγματο χάρη. Αν σκεφτούμε κάτι έναν βραστήρα που είναι στεδεμένος με υπολογιστή, είναι διαφορετικό σε μια, αν χρησιμοποιήσει το βραστήρα σε ένα νοσοκομείο στο σπίτι σου, ένα παράδειγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα και άλλα είδη κινδύνων. Ε, λοιπόν, η εφαρμογή τη διαφοροποιημένη αυτή προσέγγιση απαιτεί μια αλλαγή τη διατυπώσεω τη προτάσεω. Επίση, συνεπάγεται ε, ότι θα πρέπει να συνεργάζεται η ΕΝΗΣΑ με διάφορε κατηγορίε ε, χρηστών, εκπροσώπου των διαφόρων τομέων των χρηστών για να καθοριστεί ε, να καθοριστούν πλαίσια προστασία και να μειωθεί ο κίνδυνο διάφορε κατηγορίε χρηστών. Μια άλλη πτυχή που είναι δύσκολο να κατανοηθεί είναι πώ αποτελεσματικά μπορεί η ΕΝΗΣΑ να εστασπίσει ένα σύστημα πιστοποίηση που θα εδράζεται επί ισχυών των προτύπων και βελτίστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει, θα πρέπει να υπάρχουν σχήματα ε, ασφαλείας για διάφορα είδη χρηστών και εφαρμογών λογισμικών. Το άθρο 45 που ασχολείται με τους στόχους ασφαλείας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης έχει ένα κατάλογο απειλών και αντιμετώπιση αυτών ασφαλείας. Δεν θέλουμε να είναι εξαιρετικό, γιατί εξαιρετικό κατάλογο θα ήταν ε, κάτι άκαμπτο και δύσκολο να ενημερωθεί θα πρέπει οι τεχνικές πτυχές να αναλυφθούν περισσότερο από την ΕΝΙΣΑ. όσον αφορά το άρθρο 46, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά την για τις πιστοποίησεις όχι μόνο για τα προϊόντα αλλά και για τις υπηρεσίες ε, που θα πρέπει να έχουν, κάποιες θα πρέπει να έχουν κάποια επίπεδα με εγγύησεις βάσει συγκεκριμένων ε, πλαισίων ασφαλείας και κινδύνων, όχι γενικόλογα. Θα πρέπει να υπάρχουν προσμετρήσιμοι παράγοντε όπω το είδο του του κινδύνου για να ελαχιστοποιούνται προσωπικέ ερμηνείε των άρθρων. Όσον αφορά την ανάλυση του άρθρου 37 τη προτάσεω, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία τη διατάξεω που θα πρέπει ε, να περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα ευρωπαϊκή πιστοποίηση, Το, το α δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε προϊόντα, αλλά επίση περιλαμβάνει ε, και άλλε στοιχείε και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν σωστές, ε, κάποιες δυνατότητες προσαρμογής απρόβλεπτε συνέπειε. Λοιπόν, η ομάδα τη κυβέρνηση ασφαλεία, αναφέρεται σύνθεση. Θα επαναλάβω υπό τον κανονισμό 2012 ε, που δεν εκπροσωπείται σωστά, δεν λαμβάνει υπόψη επιτοχέ. οι Ποιε θα πρέπει να ακυρώσει δυνάμει του άρθρου 54 τη προτάσεω. Όπω γνωρίζετε, προβλέπεται ότι ένα κάτω τη Ευρωπαϊκή Ενώση μπορεί να καθορίσει διατάξει για ακυρώσει που θα πρέπει να επιβληθούν. Εφόσον εθελοντικά τα σχήματα δεν είναι σαφέ ποιο και πώ θα, επι... θα δέχεται τι κυρώσει. Μια κυρώση, κατά την άποψή μα, θα πρέπει να επιβάλλεται εάν δίνονται επιστοπίσει για προϊόντα και υπηρεσίε χωρί να πληρούνται τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφέ. Θα πρέπει να, η ΕΝΗΣΑ να μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχου, να, να εξακριβώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίε πληρούν τι προποθέσει και με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων για, που θα πρέπει να εντάσσονται συγκεκριμένα πλαίσια ασφαλεία. Και θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, οι διάφοροι αρμόδιοι φορεί. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα και το θυσιαστούμε επιθεμάτων που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ αυτή τη προτάσεω και των υφισταμένων φορέων. Επί παραδείγματι, στο άρθρο 44 αναθέτει στην ενίσα τη λειτουργία που ήδη προβλέπεται για τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς κύρωση εξαφρίβωσης. Θα πρέπει αυτή η διάταξη να διευρυνθεί ούτως ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη των στόχων μεταξύ των διαφόρων φορέων. Επιπλέον, θα πρέπει να τροποποιηθεί και αναφορά στο άρθρο 48-4 γ, όπου μόνο η ΆΖΟ, η ΑΕΤΑ αναφέρεται και τα διάφορα άλλα πρότυπα. Εάν θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα πρέπει και το 17-21 και 17-24 του ΕΑΖΟ να ληφθούν υπόψη και τα 49 για τις εθνικές πιστοποίησεις κυβερνοασφαλείας θα πρέπει να χορηγούνται με σωστή προσέγγιση να μην υπάρχει επικάλυψη και ε, αντίκρουση μεταξύ, σύγκρουση μεταξύ των φορέων. Ε, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των εθνικών φορέων ε, επικύρωσης δεν θέλουμε να υπάρχει επικάλυψη με την κίνηση των εθνικών φορέων. Το άρθρο 50 προβλέπει το διορισμό εθνική αρχή πιστοποίηση που θα πρέπει να καλύπτεται από υφιστάμενε αρχέ, να μην δημιουργηθούν νέε, για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα να ξενομήσουμε κόστο. Αλλιώ θα είναι αναπόφευκτη επικάλυψη πιστοποίησης. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού κανονισμού ε, θα πρέπει να επενεθεί. Υπό το φω όμω των ανωτέρω αναφερθέντων χρειάζονται αλλαγέ στο κείμενο και κυρίω όσον αφορά τη, μια διαφορετική προσέγγιση που θα βασίζεται στη μείωση του κινδύνου και όχι σε συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα και θα πρέπει να έχουμε και διάφορα εχέγγυα με βάση ε, τους κινδύνους και την ασφάλεια για την πιστοποίηση. Και θα πρέπει ενίσα να διεξάγει ελέγχους επί πιστοποιηθέντων προϊόντων και υπηρεσιών και θα πρέπει όμως να εμπλακούν επίσης και άλλοι φορείς των οποίων η άποψη λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Καταφέρατε μέσα σε 8 λεπτά να καλύψετε 50 παραγράφους. Μπράβο σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ηλία Χάντζο, που είναι διευθυντής για κυβερνητικές ε, υποθέσεις ε, στον όμιλο Σιμαντέκ ε, για προγράμματα στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία, Ειρηνή, Ειρηνικό και Ιαπωνία. Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο λοιπόν σε αυτό το καλεσμένο μας, στον κύριο Χάντζο, που είναι επίσης ε, αρμόδιος ε, και σύμβουλος για θέματα κρίσιμων υποδομών. Ε, μάλιστα, έχει τυχαίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπούδασε στα πλαίσια του Έρασμος στο Πανεπιστήμιο του Λίμπουργκ, έχει μεταπτυχιακό σε δίκαιο επικοινωνιών και υπολογιστών από το Queen Mary College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου, μεταπτυχιακό σε δίκηση επιχειρήσεων από το Solway Business School Επίσης, ε, ολοκλήρωσε ε, επιμόρφωση για εκτελεστικά ζητήματα στην Σχολή Δημόσιας Δίκης του Harvard, JFK. Έχει διοριστεί μέλος στην ομάδα μονίμων ενδιαφερομένων του οργανισμού ENISA, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ασφάλειας ε, των Πληροφοριών και επίσης συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοεγκλήματος της Ευρωπόλ. Πολύ πλούσια στα διαδρομία και πολύ μεστό βιογραφικό, οπότε ελπίζω να καταφέρετε και εσείς μέσα σε ένα οχτάλεπτο να ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ε, αξιότιμοι εμπειρογνώμονες, ε, ε, Ευχαριστώ τους οργανωτές για την ευκαιρία που μου έδωσαν να έρθω σήμερα και να σας μιλήσω. Άκουσα πολλούς να μιλούν για συνεργασία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, είμαι και μέλος ε, του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του ΕΝΙΣΑ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για συνεργασία με τον κλάδο ΕΝΙΣΑ. Επίσης, ε, συμμετέχω και στο ΝΑΤΟ, στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο επίσης και στο ECR, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνών Εγκλήματος και πραγματικά έχω μεγάλη πείρα από την συνεργασία που λαμβάνει η χώρα στο κλάδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το πλαίσιο πιστοποίηση, να σα πω λίγα λόγια για τον όμιλο Symantec. Για να δείτε σε αυτό το πλαίσιο τα σχόλια μα. Είμαστε μια εταιρεία λογισμικού, αλλά προσφέρουμε υπηρεσίε νεφοπολογιστική, διαχείριση, ε, συσκευέ, ε, δραστηριοποιούμαστε στην έρευνα και φυσικά σε ΣΔΙΤ, σε συμπράξει σε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιον προστατεύουμε. Κυρίως ε, ασχολούμαστε με θέματα κυβερνοασφάλειας, οπότε προστατεύουμε κυβερνήσει, κρίσιμες υποδομές, μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι από εσά θα γνωρίζετε ε, το Norton Internet Security και Technology, ένα προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και 30 χρόνια. Και ε, είναι κυρίως πολιτική εταιρεία για τα θέματα καταναλωτή και έχει προχωρήσει πολύ η θέση να αναβαθμιστεί στην αγορά. Να σας πω πώς ε, δουλεύουμε. Καταρχήν έχουμε στενή συνεργασία με πολλά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα κράτη-μέλη ε, και σε σχέση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού ε, κλάδου, αλλά και προσφορά συμβουλών σε καταναλωτές. Καταρχήν, εγώ ειδικεύομαι σε θέματα διαδικτύου των πραγμάτων, γιατί το όλο θέμα της πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας ε, ε, με τον τρόπο που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσιάστηκε στη σημασία που θα έχει το διαδίκτυο των πραγμάτων που θα αποτελέσει εκλεκτό στόχο των hacker ε, γιατί στην αγορά. Έχουμε πολλές τεχνολογίες και θα βρεθούν στο στόχαστρο των ε, εγκληματιών αναφυσβήτητα. Όλο και περισσότερες τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων έγιναν στόχος από τους hacker και στο μέλλον θα συνεχίσουν να είναι στόχος των ε, hacker γιατί τέτοιες τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων γίνονται πια πανταχού παρούσες στην, ε, στην κοινωνία μας και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε τέτοιες συσκευές για να ανταλλάξουμε πληροφορίες ε, και οι πληροφορίες είναι ισχύς, εξουσία. Κάποιες στατιστικές ε, που δείχνουν ακριβώς αυτό το, αποδεικνύουν αυτό το επιχείρημα. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε ένα ε, πολύ δημοφιλές σύστημα λειτουργικό και τέσσερα λεπτά από τη στιγμή που αρχίσαμε να λειτουργούμε γίναμε θύματα επίθεσης. Όταν είχαμε ε, το 2016 δύο λεπτά δεχτήκαμε επίθεση σε περίπτωση που ήταν απροστάτευτα τα συστήματά μας. Και αν δείτε μια γεωγραφική κατανομή τέτοιων συμβάντων κυβερνοασφάλειας ε, και στο διαδίκτυο των πραγμάτων, διαπιστώνουμε ότι γίνονται επιθέσεις ε, κυρίως στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείε, και αν προσθέσουμε τα επιμερους κρατημέλη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνουμε στο 12 περίπου το 100. Οπότε το τρίτο σημαντικό θύμα της ε, επίθεσης αυτής είναι η Ευρώπη. Και βλέπετε ότι η τάση καταδεικνύει μια νοδική πορεία του αριθμού των επιθέσεων. Οπότε σίγουρα ε, και στο διαδίκτυο των πραγμάτων η κυβερνοασφάλεια θα, γίνει, θα είναι και θα παραμείνει θέμα. Τώρα, βλέπουμε τη διαφορά της ασφάλειας μεταξύ ε, υπολογιστών, και διαδικτύων των πραγμάτων. Υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις. Ο κόσμο των διαδικτύων των πραγμάτων είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Γιατί Έχουμε το firewall και άλλους μηχανισμούς προστασίας στου προσωπικούς υπολογιστέ, ε, που ε, δεν ισχύουν για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Εκεί έχουμε ε, χιλιάδες φορείς, επιχειρησιακά συστήματα, δισεκατομμύρια προϊόντα, διαφορετικούς επεξεργαστές, οπότε υπάρχει τεράστια διαφορά. Και η ασφάλεια του διαδικτύου των πραγμάτων θα πρέπει να λάβει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ασφάλεια που εφαρμόζουμε στου υπολογιστέ. Γιατί στον κόσμο των υπολογιστών επαφιόμαστε στην ασφάλεια με βάση το, το σημείο του τελικό. Δηλαδή ε, κλειδώνοντα συγκεκριμένη συσκευή. Αυτή ιστορικά ήταν η προσέγγιση. Εδώ, για το διαδίκτυο των πραγμάτων χρειαζόμαστε μια αποκεντρωμένη ασφάλεια, κατανεμημένη σε διάφορα σημεία ελέγχου, Οπότε θα πρέπει να στηριχθούμε στην ανάλυση, στις στα συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, στην προστασία του κωδικού, του νέφους και όχι στην υπολογιστική ισχύ του συγκεκριμένη συσκευή. Βλέπετε στη διαφάνεια αυτή πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος και πόσο διαφορετικά είναι τα σημεία ελέγχου, πόσο περίπλοκη είναι η κατανομή ε, των επιμέρους χαρακτηριστικών της ασφάλειας για να είμαστε αποτελεσματική. Θα πρέπει να, στη, να προστατεύσουμε τα δεδομένα του νεφου, τις gateways και τις πληροφορίες που μπαίνουν ε, στις συσκευές, όχι μόνο τις συσκευές. Οπότε χρειάζομαστε μια πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας. Νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έργο σε επιμέρους ε, ε, τμήματα, σε ό,τι φορά τα καταναλωτικά αγαθά, τα παροχημένα συστήματα ή κάποιες ιδιαίτερες τεχνολογίες, ε, ε, προϊόντα που σχεδιάζονται χωρίς ε, εσωματωμένη ασφάλεια. Βλέπετε λοιπόν, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσβλέπουμε στο ίδιο, στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο στόχο ασφάλειας που έχουμε για τους υπολογιστές και να το αναμένουμε κάτι τέτοιο από το διαδίκτυο των πραγμάτων. Ε, τώρα το προαιρετικό σύστημα, η προαιρετική παστοποίηση θα λειτουργήσει. Ναι, αλλά χρειάζεται να υπάρχει αγορά για κάτι τέτοιο, εναρμονισμένη. Και επίση θα πρέπει η ενιαία αγορά να λειτουργεί εδώ. Και φυσικά να είναι απαραγμένο από τη γραφειοκρατία ένα τέτοιο προαιρετικό σύστημα. Οδεύουμε προς σωστή κατεύθυνση. Έχω κάποιε επιφυλάξει. Ε, καταρχήν, βλέποντα πω συνεχίζονται οι συζητήσει για την ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων, τι να σας πω, χρειαζόμαστε πάντως μια ξεκάθαρη άποψη για το τι θα πιστοποιηθεί, πού και ποιος θα είναι ο ρόλος των επιμέρους φορέων. Γιατί ε, άλλο ρόλο θα έχουν οι κατασκευαστές ε, ηλισμικού και άλλο ρόλο οι κατασκευαστές ε, λογισμικού ή πάροχοι δικτύων. Επίσης, ε, η ασφάλεια του διαδικτύου των πραγμάτων δεν θα λειτουργήσει με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει να είναι μεγάλη κλίμακο, ε, να είναι αυτοματοποιημένη διαχείριση των δικτύων και επίση ε, να καθοδηγείται από την αγορά, ε, να προσαρμόζεται στην αγορά αν υπάρχουν ικανότητες που θα συνδέονται με αυτή την πιστοποίηση και επίσης να είναι πανευρωπαϊκή, να μην στηρίζεται σε εθνικά μοντέλα. Επίσης θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι, να συμμετέχει και ο ιδιωτικός κλάδος ε, στην ε, θέσπιση του και κάποιοι ε, κανονισμοί που υπάρχουν όπως το η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και φυσικά σημαντικός ρόλος και του οργανισμού ΕΝΙΣΑ. Ευχαριστώ και με στη διάθεση να απαντήσω σε ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και εσείς ε, ε, σεβαστήκατε το όριο των 8 λεπτών και μπράβο σας. Να συνεχίσουμε τώρα με τις τοποθετήσεις σας. Κάθε εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας θα έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του. Στον δεύτερο γύρο, όποιος επιθυμεί να προβεί σε τοποθέτηση, θα λάβει χρόνο ενός λεπτού. Πρώτη η κυρία Νίπλερ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε το λόγο κυρία Νίπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο προσκεκλημένους του δεύτερου γύρου για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, τοποθετήσεις. Έχω τρεις ερωτήσεις. Θέλω πρώτα να ρωτήσω εάν χρειαζόμαστε οικειοθελέ ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποιήσεων ή υποχρεωτικό. Αυτό θέλω να μάθω από τον κύριο Χάντζο άκουσα ότι αρκεί οικειοθελέ σύστημα εφόσον υπάρχει αγορά. Υπάρχει ήδη αυτή η αγορά, αυτή είναι η ερώτησή μου τώρα. Ή πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η αγορά. Το λέω έτσι κάπως απλουστευτικά. Εμείς... Αν θέλει να μου απαντήσει εάν ποια θα, θα πρέπει να είναι τα κίνητρα για να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε αυτό το οικειοθελέ σύστημα. Δεύτερο, Χρειαζόμαστε προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, στην ανάλυση του κινδύνου. Ε, δεν γνωρίζω τόσο καλά τα πράγματα. Όμως νομίζω ότι είναι διαφορετική η βαρύτητα των κινδύνων εκάστοτε και θα πρέπει η πιστοποίηση να υπακούει σε ένα αντίστοιχο κριτήριο. Τρίτο, μπορεί η πιστοποίηση να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Τι γίνεται με τις ΗΠΑ και με την Κίνα, έχουν τέτοιε πιστοποίησεις, έχουν τη δυνατότητα να υπαγορεύσουν τα διεθνή πρότυπα ή μπορούμε εμείς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα να ηγηθούμε και να τα υπαγορεύσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ κύριε Νίπλε, ο πρόεδρος κύριος Κόχλιτσεκ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Άλμπρεχτ, τον οποίο καλωσορίζω κιόλα. Είναι εκπροσωπή εδώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ Προστασίας Καταναλωτών. Από τη σκοπιά της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Πρώτα, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Νίπλερ, που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο σημαντικό ερώτημα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού ενίσα. Αν θα πρέπει δηλαδή το σύστημα πιστοποίησης να είναι και ο θελές υποχρεωτικό. Βεβαίως διαστρωματώνεται κάπως η ερώτηση, διότι τι σημαίνει υποχρεωτικό, δεσμευτικό, binding, θα είναι ο μοναδικός τρόπος πιστοποίησης ή θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν πράγματι διαφορετικές, διαφορετικά στρώματα. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το ερώτημα προχωρούμε προς την κατεύθυνση προτύπων της ευρωπαϊκής αγοράς σε κάποιο βαθμό, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ασφάλεια της πληροφορικής. Και η εντύπωση που έχω, αλλά και οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, είναι ότι εάν επιθυμεί κανείς να φτάσει σε κάποια πρότυπα στην κοινή αγορά κάποιου είδους δεσμευτικός μηχανισμός θα πρέπει να θεσπιστεί γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θεωρούμε ότι μας επιτρέπει να επιτύχουμε κοινά πρότυπα. Θα ήθελα ωστόσο να ακούσω την άποψή σας για, για αυτό το θέμα, το οποίο το θεωρούμε κλειδί. Ευχαριστώ ερώτηση της δεσμευτικότητας ή έστω μέρους του συστήματος πιστοποίησεως είναι σημαντική και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη και των δύο ομιλητών. Εκ μέρους της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Κουρουμπάσεφ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω στο ερώτημα αν θα είναι δεσμευτική ή δεσμευτικός, δεσμευτικό ή και ο το σύστημα. Έχω ακούσει απόψεις και τα δύο. Η νομοθεσια ή e-privacy είχε προκαλέσει τέτοιες συζητήσεις. Θυμάστε την μη δεσμευτική πιστοποίηση των τελικών συσκευών. Και κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε είναι αν θα πρέπει να μιλούμε για επίπεδα πιστοποίησεως στην παρούσα νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χαμηλότερο επίπεδο πιστοποίησεως για καταναλωτές, ένα δεύτερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις ή τη βιομηχανία και ένα τρίτο επίπεδο για κυβερνητικά όργανα, υπουργεία και ούτω καθεξής. Άρα, ε, τρία διαφορετικά επίπεδα. Και ένα άλλο ζήτημα που συζητήσαμε συστήματα εθνικής ή μάλλον εθνικά συστήματα πιστοποίησης, γιατί υπάρχουν τέτοια. Εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης, τι θα γίνει με τα εθνικά, μπορούν να συνεπάρχουν τα εθνικά. Και για την ανταλλαγή πληροφοριών αυτή γίνεται στο διακρατικό επίπεδο. να υπάρχει σύστημα πιστοποίησης που θα εκδίδει πιστοποιητικά τα οποία θα μπορούν να ξεπερνούν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούν να ισχύσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος Κόχλητσα και είναι σημαντικό όντως να διακρίνει κανείς ανάμεσα στην πιστοποίηση Ενό απλού προσωπικού υπολογιστή και ενό πυρηνικού εργοστασίου. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαφορά. Ο κύριος Κοσινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να πω κάτι βασισμένο σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Έχω μία ερώτηση. Τι πρέπει να πιστοποιήσουμε. Διότι στον εμπορικό τομέα υποστηρίζουμε η πιστοποίηση αφορά ένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Παράδειγμα αυτού είναι η Symantec. Έχουν βασίσει την επιχείρησή τους επ' αυτού, δηλαδή την προστασία από τους ιούς κλπ. Αυτό που ανέφεραν οι συνάδελφοι αφορά και κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να κάνουμε διαφοροποίηση από το δημόσιο τομέα της πιστοποίησης χωρίς να αυξήσουμε το γραφειοκρατικό άχθος μέσω των διαδικασιών αυτών. Και, και, πού πρέπει να υπάρχει διεθνής πιστοποίηση και πού πρέπει να εφαρμόζουμε ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Εδώ μιλάμε για μεγάλα ποσά. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Κάτι έλειπε. Η διανομή των πληροφοριών, η διαβίβαση πληροφοριών προς το κοινό ούτως ώστε ο κόσμος να μην βασίζεται πολύ λόγω ελλείψεως γνώσεων σε λάθος σύστημα προστασίας. Να πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι κάποια συστήματα μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Ότι όταν συνδέεσαι με το διαδίκτυο δεν έχει κάποιους κινδύνους. Όταν δεν έχει προστασία. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη πρέπει καταναλωτών, να φυλάγονται κάπως. Χρειάζεται αύξηση της ευαισθητοποίησης, αυτό είναι σημαντικό και δεν είμαι σίγουρος αν αυτό έχει γίνει πρόσφατα στο κατάλληλο επίπεδο να καταλάβει ο κόσμος. Πιστεύετε ότι έχει γίνει αυτό είναι μια ερώτηση και ευχαριστώ πολύ και για τα παραδείγματα που αναφέρατε. Και τώρα ο εκπρόσωπος της Άλτα. Η... Ε, ε, κυρία Κάλλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ερώτηση για τον τελευταίο εμπειρογνώμονα. Στη διαφάνεια αναφέρθηκε στα συστήματα πιστοποίησεως. Και είπατε ότι ο κανονισμός περί ιδιωτικότητας Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Ήμουν εισηγήτρια για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα στην Επιτροπή. Αφήσαμε την πτυχή εκτός, διότι ξέραμε ότι έρχεται η δέσμη μέτρων για την κυβερνοασφάλεια. Άρα δεν υπήρχε νόημα να γίνει επικάλυψη. Μήπως μπορείτε να δώσετε λεπτομέρειες. Έχετε άλλε ανησυχίε που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και το σχετικό κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και αυτό σε συνάρτηση με την κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή, πολύ σχετική ερώτηση. Υπάρχει κάποιο εκτό του κυρίου Άλμπρεχτ, υπάρχει άλλο εκπρόσωπο των Πρασίνων που θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Η ε, Τιγκού είμαι εγώ. Η FTD. Υπάρχει κάποιος από το FTT που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι. Η ΕΝΕΦ, η Κρίστα Λεβασχία φύγε. Δεύτερος γύρος λοιπόν. Ο κύριος Ρούμπικ, συνάδελφε Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για όλους μας είναι το θέμα ενδιαφέρον διότι πρόκειται για τα πλαίσια που θα ισχύσουν στο μέλλον. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σύστημα ΣΤΟΑ της αξιολόγησης τεχνικών επιλογών. Έχει αναθέσει μελέτη. Με τη μελέτη αυτή νομίζω θα φανεί που βρίσκονται και τα προβλήματα. Και θα πρέπει να γίνει και κατηγοριοποίηση των πιστοποίησεων hardware, software κλπ. Θέλουμε να γνωρίζουμε επίσης ποιοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται, πού χρησιμοποιείται η τεχνητή ευφυΐα. Είναι σημαντικό και για τον τελικό καταναλωτή να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Νομίζετε ότι τα συστήματα πιστοποιήσεως όπως ο TÜV για παράδειγμα μπορεί να συστήνει στους καταναλωτές ότι θα πρέπει να αγοράζει μόνο τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν και την τελική πιστοποίηση. Υπάρχουν και πολλά περιοδικά τα οποία τα δείχνουν αυτά και μάλιστα διαφανώς. Ευχαριστώ, πράγματι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, λέει ο πρόεδρος Κοχλίτσεκ. Υπάρχει άλλος κανείς ο οποίος ε, θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο για το θέμα. Κανείς, καλώς. Άρα ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Φατζόλη και στον κύριο Χάντζο για πέντε λεπτά στον καθένα για να μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Κύριε Φατζόλη, εσείς πρώτος. Ευχαριστώ. Απαντώ Ιταλιστή. Και θα πάω πιο σιγά, έτσι θα μιλήσω πιο αργά από ό,τι πριν. Πρέπει να είναι κάτι υποχρεωτικό, όχι. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια πλαίσια της αγοράς που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο, ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως κρίσιμες υποδομές, τραπεζικός κόσμος, τομέα της υγείας. Υπάρχουν απαιτήσει όσον αφορά την πιστοποίηση, διότι είναι προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιηθούν και μπορούν να έχουν αντίκτυπο επί της υγείας των πολιτών και επί της ασφάλειας των πολιτών. Μετά στρέφομαι στην τρίτη ερώτηση όσον αφορά την προσέγγιση που εδράζεται επί του κινδύνου, για να γίνω σαφέστερος. Η θέση μας είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η πιστοποίηση. Από την άλλη πλευρά όμω δεν θα πρέπει να γίνει ένα στοιχείο που να στρεβλώνει την αγορά. Είναι προφανέ λοιπόν ότι μια πτυχή της πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν ακολουθεί την καθημερινό κατακαιρματισμό με κόστος που συνεπάγεται αυτό αλλά προσθέτει αξία, κάτι τέτοιο είναι σίγουρος ε, ο δρόμος που να ακολουθηθεί. Η άλλη ερώτηση, αν υπάρχει αγορά, μια αγορά που μπορεί να έχει η δική του αξία. Εμείς πιστεύουμε ότι σίγουρα ναι, η αντίληψη που έχουμε και σαν ένωση και σαν ε, αρχή ε, που ε, εκπροσωπούμε το δημόσιο τομέα και τις εταιρείες και τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, και μας λένε κατά πολύ όλοι αυτοί που εκπροσωπούμε ότι αυτό έχουν απέτηση ησυχία όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσία που διατίθενται και αυτό ε, δημιουργεί ε, οι ασφαλές υπηρεσίες και προϊόντα ανοίγουν μια αγορά. Έχουμε διάφορες, ε, διάφορα αιτήματα για περισσότερη ησυχία και ηρεμία όσον αφορά τον εφοϋπολογιστικό τομέα, cloud computing. Και εκεί χρειάζεται αυτό. Και μετά η προσέγγιση που βασίζεται από του κινδύνου. Εμείς είμαστε απόλυτα πεπισμένοι γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν πρέπει να λάβουν υπόψη, ε, υπάρχει ένα λογαριασμό, άλλο λογαριασμό σε έναν προσωπικό υπολογιστή και άλλο σε πυρηνικό υπολογιστή. Ένα λογαριασμό χρησιμοποιείται, παραδείγματο χάρη στο σπίτι μου, και ένα άλλο σε ένα πυρηνικό, ε, πυρηνική μονάδα. Δηλαδή, πιστοποίηση για ένα προϊόν που χρησιμοποιώ για οικιακού σκοπού είναι άλλο πιστοποιητικό από το ίδιο προϊόν που μπορεί να είναι ίδιο, ο ίδιο υπολογιστή χρησιμοποιείται όμω σε πυρηνικό αντιδραστήρα και μπορεί εκεί ε, να έχει και ένα σύστημα προσωπικών υπολογιστών ή συστήματα ε, με κάμερες και βίντεο παρακολούθηση που χρησιμοποιούν αυτά τα μηχανήματα. Και μπορούν να γίνουν επιθέσεις. Άρα θα πρέπει να, να έχουμε, να υπόψη και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του μηχανήματος και πού χρησιμοποιείται. Και ποιο διαδρομή πρέπει να ακολουθήσουμε για την επιστοποίηση. Η επιστοποίηση θα πρέπει να εδράζεται βασικά επί της χρήσεως του προϊόντος και της υπηρεσίας και βάσει αυτού μετά να γίνεται αξιολόγηστη ε, ποιε είναι οι ανάγκες και οι προποθέσει για την πιστοποίηση και ποιο είναι το πλαίσιο πιστοποίηση που πρέπει να δημιουργήσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ και, και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ο γιος Χάντζος, που θα μπορέσει να τοποθετεί ως τελευταίο εμπειρογνώμων. Πολλέ ερωτήσει, λίγο δύσκολο να τι συμπιέσει κανεί όλε, θα για να τι απαντήσει το δυνατόν ταχύτερα, αλλά φαίνεται να συγχέουμε ωστόσο στη συζήτηση τρία διαφορετικά πράγματα. Πιστοποίηση που είναι ένα ξεχωριστό πράγμα, έχει ιδιαίτερη σημασία, τις μακροπρόθεσμες ανάγκε ανάγκες ασφαλείας, άλλο ξεχωριστό αυτό, και τέλος την επισήμαση, το labeling. Άκουσα να μιλούν κάποιοι από εσά για την awareness, τη συνειδητοποίηση. Αυτό όμως δεν είναι ζήτημα της πιστοποίησης. Εκεί βάζετε απλώς ένα χ σε ένα κουτάκι. Το labeling θα σας δώσει την συνειδητοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηχάνημα, ε, συνδέεται με το ΑΒΓ δίκτυο και έχει τα εξή χαρακτηριστικά ασφαλείας. Έλληνας είμαι, μου αρέσουν τα ιστορικά. Αν εξετάσετε την ιστορία, θα, σας, δείτε ότι μας διδάσκει η ιστορία ότι έχουμε συστήματα πιστοποίησης, τα κοινά κριτήρια, είναι τα οποία, τα οποία μάλιστα είναι πολύ όριμα. Ποιος τα χρησιμοποιεί? Μόνο ο στρατός και μόνο ο στρατός διότι χρειάζονται αυτό το επίπεδο διασφάλισης και καμιά φορά ούτε και τους ίδιους στρατιωτικούς δεν τους ικανοποιούν διότι σημαίνει ότι είναι άκαμπτο το σύστημα και δύσκολο να αλλάξει. Φανταστείτε να πιστοποιήσετε μια ιατρική συσκευή σε υψηλό επίπεδο, που είναι πραγματικά σημαντικό και αναγκαίο. Αυτό σημαίνει όμω ότι δεν μπορείτε να το αγγίξετε. και μπορεί να έχετε σχετικέ εμπειρίε που να δείχνουν ότι πρέπει να κάνετε κάποια αλλαγή. Έχουμε πιστοποίηση για κάποια συσκευή και στο επίπεδο αυτό δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Άρα δεν μπορούμε και να την επικαιροποιήσουμε, γιατί τότε δεν μπορούμε να την πιστοποιήσουμε πάλι. Αυτά είναι κάποια από τα πρακτικά ζητήματα που θα προκύψουν. Τι σημαίνει πιστοποίηση και σε ό,τι αφορά το κόστο. Αν μιλούμε για εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι φανταστικά τα νούμερα αυτά για να πιστοποιηθούν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα και η Symantec έχει για παράδειγμα 200 προϊόντα. 200 εκατομμύρια δολάρια Ποιο, η ευρώ, ποιος θα πληρώσει αυτά. Και τι πάει να πει για την ανταγωνιστικότητα μια μικρομεσαίας επιχείρηση εάν αυτά που θέλετε, αυτό που θέλετε να πετύχετε είναι πράγματι η Ευρωπαϊκή ενιαία Αγορά. Χρειαζόμαστε μια risk-based approach. Μάλιστα, βεβαίω. Γι' αυτό εξασέριξα τη διαφάνεια με τα διάφορα πράγματα και τα διάφορα επίπεδα ασφάλεια. Δεν μπορείτε να αναμένετε να εξασφαλίσετε με τον ίδιο τρόπο μια απλούστατη συσκευή, μια κάμερα για παράδειγμα, η οποία δεν έχει καν και ε, επεξεργαστεί με τον ίδιο τρόπο που θα επιστοποιήσετε το, τη, την καρδιά ενός πυρηνικού σταθμού. Εκειοθελές λοιπόν το σύστημα. Ναι, αυτό θεωρούμε, διότι η ε, οδηγία NIS προβλέπει τη σχετική βάση. Τίθεται το ερώτημα, πώς δημιουργείται τα κίνητρα μέσω της αγοράς, ώστε να θέλει ο κόσμος να προχωρήσει στην πιστοποίηση. Συγκεκριμένο παράδειγμα, σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμε και δραστηριοποιούμε σε πολλές. Η συζήτηση είναι σχετική με το GDPR. Πολλοί πελάτες έρχονται και μας λένε δώστε μου το επίπεδο διαβεβαίωσης που χρειάζομαι για το GDPR. Ο οργανισμός που θα σου δώσει το διεθνές αυτό οργανισμένο ε, πιστοποιητικό θα λάβει τα χρήματα τελικά. Διότι όλοι μας θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής, επαρκές κίνητρο από την αγορά. Θα χρειαστεί λοιπόν να βασιστούμε στην αγορά. Η αγορά θα οθήσει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και όχι ο νομοθέτης που θα τα γράψει σε πέτρα. Ελπίζω ότι απάντησα για το οικειοθελές ή δεσμευτικό. Εγώ θα ήθελα ένα μη δεσμευτικό σύστημα το οποίο θα το στηρίξει η αγορά. Risk-based approach. Η Κίνα έχει καθεστώς πιστοποίησης. Ναι, οι διεθνείς παίκτες προσπαθούν να συμμορφωθούν με το σύστημα αυτό πολλοί από τους διεθνείς παίκτες και Ευρωπαίοι κιόλα έχουν πολύ σημαντικές ανησυχίες σχετικά με το ζήτημα εμπιστοσύνης που έχει σχέση με αυτό το σύστημα πιστοποίησης και το λαμβάνουν υπόψη. Προφανώς εάν καταλήξουμε σε πιστοποίηση και μιλούμε τότε για διαφορετικά επίπεδα, ναι. Και εάν ακολουθήσουμε την οδό της πιστοποίησης για να υιοθετηθεί από την αγορά θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκό. Δεν έχει κανένα νόημα να είναι διαφορετικό για τη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Πορτογαλία. Για την κυρία Κάλλας, για την e-privacy. Οι ανησυχίες που έχει εκφράσει ο κλάδος της ασφάλειας αναφέρεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8. Πρόσβαση σε τελικές συσκευές χρήσης και επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς κυβερνοασφάλειας διότι πρέπει να μπορούν να διασυνδέουν τις πληροφορίες σε ένα περιβάλλον προστασίας του διαδικτύου των πραγμάτων. Είναι σωστό δηλαδή αυτό που είπατε, αλλά υπάρχουν και άλλες ανησυχίες. Προσπάθησα να απαντήσω όλα μέσα σε πέντε λεπτά, αγαπητέ Πρόεδρε. Μάλιστα, θαυμάσια. Τώρα θα ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Δέσποινα Σπανού, που είχε ήδη ξεκινήσει να απαντά και για τις ερωτήσεις του δεύτερου σκέλους της δημόσιας ακρόσης. Αν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Καταρχήν για το ρόλο του ΕΝΙΣΑ στα πλαίσια της πιστοποίησης. Να πούμε δύο λόγια για τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Η πρόταση προβλέπει ένα σύστημα προαιρετικής πιστοποίησης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες να λαμβάνουν πιστοποίηση. Οπότε ξεκινάμε αυτό το πρώτο βήμα της εθελοντικής πιστοποίησης, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το σύνολο της αγοράς της κυβερνοασφάλειας. Η ιδέα είναι η αγορά από μόνη της να αποφασίσει πού χρειαζόμαστε κατά προτεραιότητα την κυβερνοασφάλεια και εκεί θα αναπτυχθούν τέτοια συστήματα πιστοποίησης. Η ιδέα ενός πλαισίου που θα επιτρέψει την έγκριση των διαφόρων μέρους συστημάτων προϋποθέτει ακριβώς την ελαστικότητα, την ευελιξία. Και το ότι το έχουμε προαιρετικό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ε, εφαρμόσιμα συστήματα. Καταρχήν, από τη στιγμή που θα εγκριθεί το σύστημα με μια εφαρμοστική πράξη θα πρέπει να ε, τύχη εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές και άρα να εφαρμοστεί, γιατί θέλουμε συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού. Ένα σύστημα δηλαδή όπου το πιστοποιητικό θα εφαρμόζεται, θα μπορεί να αμφισβητείται αν δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και ούτω καθεξής. Παρά την προαιρετικότητα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά πιστοποιητικά που ρωτήσατε, με βάση την πρότασή μας, από τη στιγμή που υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα, τα εθνικά πιστοποιητικά για το ίδιο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών καταργούνται από τη στιγμή που θα φτάσουν στην ημερομηνία εκπνοής τους. Θέλουμε κάποια ασφάλεια στην αγορά και να αποφύγουμε την επικάλυψη ακριβώς. Αυτή την επικάλυψη θέλουμε να αποφύγουμε στην πρόταση. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα επίπεδα διαβεβαίωσης, η πρόταση, όπως είπατε, προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα διαβεβαίωσης. Και τέλος, για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Τα προτινόμενα συστήματα που θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν με βάση τη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης ε, δεν αποκλείεται να μεταξελιχθούν σε πλήρως ανεπτυγμένα δημόσια πρότυπα. Οπότε μπορεί να έχουμε μια αγορά στην Ευρώπη που θα συγκλίνει με τη διεθνή αγορά, ακριβώς γιατί πραγματικά αν υπάρχουν τέτοιες διεθνείς προδιαγραφές ή διεθνή πρότυπα για τέτοια προϊόντα υπηρεσίες, αυτά θα γίνουν τα σημεία αναφορά σε πολλές δικαιοδοσίες. Και μάλιστα πολλέ δικαιοδοσίε ανά τον κόσμο εξέφρασαν ενδιαφέρον για την πρόταση επιστοποίηση που κάναμε, ακριβώ για αυτό το λόγο, γιατί προβλέπει την ευελιξία. Και ελπίζω να κάλυψα όλε τι ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Σπανού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά που μπόρεσα να προεδρεύσω σε αυτό το τμήμα της ακρόασης και να ευχαριστήσω θερμά και του συναδέλφου που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και κυρίως την κυρία Σπανού που μας έκανε μια εισαγωγή στον τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε υπόψη στις δικές μας εργασίες. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Έχουμε κερδίσει και 8 λεπτά οπότε αν δεν έχετε αντίρρηση και δεν ακούσα διαμαρτυρίες θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο, πολύ σημαντικό και θα μας το παρουσιάσει η κυρία Αγγέλικα Νίμπλερ. Οπότε αφήνω τους καλεσμένους μας, τους εξέχοντες καλεσμένους μας, ε, λίγα δευτερόλεπτα να αποχωρήσουν από την αίθουσα και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Νίμπλερ για να μας ενημερώσει για την αποστολή της Επιτροπής στον ΕΝΙΣΑ. Συνεχίζει ο, ο πρόεδρος Κόλιτσεκ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε επιτροπή έστειλε μια αντιπροσωπεία δύο προσώπων στον οργανισμό ΕΝΙΣΑ στην Αθήνα 19 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 Θα αφιερώσουμε λοιπόν πέντε λεπτά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το πιο σημαντικό είναι η κυρία Νίμπλερ να μας ενημερώσει σχετικά με τις εντυπώσεις της από την ε, αντιπροσωπή αυτή από την αποστολή μάλλον αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Πράγματι δεν νομίζω να χρειάζομαι και περισσότερα από πέντε λεπτά. Πήγαμε την κυρία Βαν Νέβενχόιζεν για δύο ημέρες στην Αθήνα, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του οργανισμού ΕΝΙΣΑ. Γνωρίζετε ότι ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε έχουμε βρει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας του διαδικτύου και επομένως με τα καθήκοντα του ΕΝΙΣΑ και τακτικά κάθε δύο χρόνια κάνουμε αποστολές στον οργανισμό αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΕΝΙΣΑ, τον καθηγητή κ. Χέμπρεχτ. Συζητήσαμε με τον επικεφαλής επιχειρησιακής ασφάλειας, κ. Δημοσθένη Οικονόμου. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής του γραφείου κ. Ράιαν και είχαμε και την ωραία ευκαιρία να συνομιλήσουμε με συνεργάτες του ΕΝΙΣΑ. Έγινε ένα είδος συνέλευσης του προσωπικού που συγκάλεσαν και μπορέσαμε να θέσουμε ερωτήσεις, μπορούσαμε, μπορέσαμε να εξηγήσουμε και την, τις πολιτικές μας προσεγγίσεις ως Επιτροπή Ήτρε. Οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από τρία βασικά θέματα, μιας και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε μόλις δει το φως της δημοσιότητας, είχαμε ενημερωθεί σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα και awareness raising του ΕΝΙΣΑ. Μιλήσαμε και το θέμα, για το θέμα cryptocurrencies, θέμα το οποίο γνωρίζει καλύτερα η κυρία Βανιούεν Χάιζεν και το συζητεί στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα είμαι σύντομος οι εντυπωσει μας. Η συνάδελφος μου Κούρα Πανιούεν Χάιζεν και εγώ συναποκομίσαμε μια θετική εντύπωση από τον οργανισμό και από άποψη προσωπικού είναι καλά στελεχωμένη η υπηρεσία αυτή. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν και ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον οργανισμό ΕΝΙΣΑ. Είχαμε και την μεγάλη ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε μια παρουσίαση για το πόσο εύκολα μπορεί ένας hacker να παρέμβει σε ένα κινητό τηλέφωνο. Είδαμε δηλαδή με πόση άνεση μπορούν να μπουν ε, στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο προσωπικό σας υπολογιστή. Είχαμε και το θέμα blockchain και κρυπτονομίσματα, το οποίο συζητήσαμε με το προσωπικό του ΕΝΙΣΑ και ευρύτερα για προστασία δεδομένων ή privacy κλπ. Ευχαρίστως εάν επιθυμείτε, ε, να φωτίσω περισσότερο πτυχές της επίσκεψής μας, αλλά συνολικά για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη και ιδίω βέβαια για ζητήματα κυβερνοασφάλειας ήταν και το σωστό χρονικό σημείο ότι πήγαμε στον Ενίσα στην Αθήνα. Ο Ενίσα μέσα από τα χρόνια λειτουργίας του έχει συγκεντρώσει πολλή τεχνογνωσία μας έδειξαν οι αρμόδιοι πόσο στενά συνεργάζονται και με τις εθνικές αρχές προστασίας και νομίζω ότι μπορώ να πω ολοκληρώνοντας ότι πρόκειται για μια ε, πραγματικά επαγγελματική απόδοση των προσπαθειών του προσωπικού που ικανοποιεί και την εντολή του και δικαιολογεί και τους πόρους του και προσωπικούς και χρηματοδοτικούς. Θεωρώ ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο οργανισμός αυτός και από εμά και στη συζήτηση τώρα για την νομοθεσία περί κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον οργανισμό και συστήνω τους συναδέλφους μου με κάποια ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη των Αθηνών. Μάλιστα ήμασταν ε, τέλη Σεπτεμβρίου και έφυγα από το Μόναχο με κρύο και έφτασα εκεί με 33 βαθμούς. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο μας συνόδευσε. Πραγματικά ήταν λοιπόν πάρα πολύ θετικέ εντυπώσεις. Δύο ημέρες μόνο, αλλά θα πω σε όλες και όλους τους συναδέλφους μου, πηγαίνετε να δείτε τον οργανισμό αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο όγκος τεχνογνωσίας που έχουν συγκεντρώσει τα μέλη του προσωπικού του ΕΝΙΣΑ μέσα στα λίγα χρόνια τη λειτουργία. του. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις από άλλους συναδέλφους ή επιθυμείτε να θέσετε ερωτήσεις στην κυρία Νίπλερ. Ο κύριος Κέρι. Κέλλη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η επιθυμειτε να θεσετε ερωτησεις στην κυρια νιπλερ ο κερι ευχαριστω πολυ προεδρε η και μας εκπροσώπησε στην ΕΝΙΣΑ και σίγουρα απόλαυσε και τη ζέστη στην Αθήνα. Αλλά δεν θα είχε πολύ χρόνο. Έχουν πολλή δουλειά αυτές οι αποστολές. Ε, αυτοί που συνάντησες, Αγγελικά, είχαν κάποιες ε, αιτήσει, προτείναν κάτι σχετικά με τι μπορεί να κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πόρους κλπ. και ποια η πρότασή τους, η άποψή τους για τον κανονισμό, για την ψηφιακή προστασία και για την ιδιωτικότητα. Υπάρχουν κενά, τα προτείναμε σωστά. Ποια είναι η άποψή τους. Μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τους hacker και αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, τέλος πάντων μπορούμε να έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι πάντα θα προηγούμεθα και ότι θα ελέγχουμε τις καταστάσεις. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, Αγγέλικα. Ευχαριστώ, ρε Πρόεδρος, για τα σχόλιά σας. Όλοι θα χαιρόμασταν αν επισκεπτόμασταν την Αθήνα για να συζητήσουμε με αυτούς τους ε, νέους. Όχι μόνο για να πάμε στην πλατεία Ομονίας και άλλα αξιοθέατα, στους επτά λόφους Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα θέλατε να απαντήσετε στον κύριο Κάρι, μήπως έχει το λόγο. Ε, ε, η Αγγέλικα Νίπλερ, δεν προλάβαμε βέβαια να δούμε τα αξιοθέατα μέσα σε δύο ημέρες με συμπεριλαμβανομένη στις αναχωρήσεις και αφήξεως δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό που είδα ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον οργανισμό ενίσα στην Αθήνα είναι να βρει πραγματικά ανθρώπους με τα αναγκαία προσόντα και δεξιότητες. Γιατί βεβαίως υπάρχει τεράστια ζήτηση για τέτοια πρόσωπα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ε, εξαρτάται και από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός χρηματοδοτικά και ε, οικονομικά καλύτερα. Αυτό σημείωσα λοιπόν από, τα, από τις πληροφορίες που μας έδωσε ο οργανισμός. Δεν είχαν πολλές επιθυμίες να εκφράσουν. Ήθελαν να προβάλλουμε το έργο του οργανισμού ΕΝΙΣΑ, να μας ε, ενημερώσουν ότι κάνουν ασκήσεις σχετικά, ότι συμβάλλουν έτσι στην συνειδητοποίηση, σε αυτό το awareness raising για τις δραστηριότητες προστασίας ε, της ε, ασφάλειας των, του διαδικτύου, αλλά Ξανά το μήνυμά τους ήταν ότι δυσκολεύονται να βρουν ικανό προσωπικό. Εάν γίνει ελκυστικός ως εργοδότης ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ, τότε βέβαια θα προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους με τα αναγκαία προσόντα. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, αυτός τους ικανοποιεί, παρακολουθούν βεβαίως προσεκτικά την εφαρμογή του κανονισμού στις ε, χώρες μέλη και υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτή του σύνεγγης, αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες που δρούν στο διαδίκτυο, τους hackers κλπ. Όμως αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς. Απλώς η φιλοδοξία τους είναι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό να το πράξουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κανείς ρεαλιστής πράγματι και να το εξετάσει ρεαλιστικά. Σημειώνω πάντως ότι ο οργανισμός τα όσα έχει ήδη επιτύχει είναι πολύ σημαντικά και πολύ στέρεα. Και βέβαια δεν είναι μόνο νεαροί άνθρωποι στις τάξεις του. Υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες οι οποίοι έχουν συλλέξει επί έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σημαντικότατο όγκο τεχνογνωσίας και αυτή η διάδραση ε, πλέον πιο όριμων ε, συνεργατών και πιο νέων συνεργατών είναι αυτή η οποία έχει διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο δραστηριότητα του οργανισμού. Είμαι βέβαιος ότι εάν ενισχυθεί και άλλο το προσωπικό του οργανισμού θα μπορέσουν, πρώτα πρώτα αν ενισχυθούν οι πόροι του οργανισμού θα μπορέσει να προσελκύσει και περισσότερο ικανό προσωπικό. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος ε, Κόκλιτσα και ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, γιατί είναι 5 και 5 ακριβώς και θα περάσουμε στη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, συναδελφοί, ότι το ελόγω θέμα είναι νομοθετική προτεραιότητα και για τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Έχουμε προβλέψει μία ώρα για τη συζήτηση της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης της κυρίας Γκροστέτ. Θα ακούσουμε πρώτα την ομιλία της ηγετριάς μας, που θα μας ενημερώσει για ένα πεντάλεπτο για το περιεχόμενο του σχέδιου έκθεσής του. Θα μας παρουσιάσει τις αδρές γραμμές της ε, έκθεσης. Μετά θα ακούσουμε για δύο λεπτά τον κάθε σκιώδη εισηγητή και τους υπόλοιπους βουλευτές στη συνέχεια για ένα λεπτό. Θα ολοκληρώσουμε με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία Γκροστέτ που θα μας ε, ανακεφαλαιώσει τη συζήτηση και τις εντυπώσεις που αποκόμισε από αυτή. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κυρία Γκροστέτα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω καταρχήν στους συναδέλφους ότι πριν από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε το σχέδιο, Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα προκειμένου να σπίσει κάποια μέτρα για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα άμυνα και ταυτόχρονα να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου της Άμυνα, τη αμυντική Βιομηχανία. Και μία από τις εμβληματικέ προτάσεις αυτού του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσεως για την ε, άμυνα είναι η σύσταση ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα για να βοηθήσει τις επενδύσεις στην κοινή έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών αμυντικών. Δύο είναι τα σκέλη. Το πρώτο σκέλος επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση συνεργατικής έρευνας, που ήδη έχουν, ε, προπαρασκευαστικές δράσεις έχουν ξεκινήσει, και το δεύτερο σκέλος στοχεύει στην απόκτηση αμυντικών δυνατοτήτων. 500 ε, εκατομμύρια ευρώ συνολικά προβλέπονται για, την περίοδο, για τη διετία 2019-2020 για να αναπτυχθούν από κοινού ε, τεχνολογίες άμυνας. 20% ε, ε, θα είναι το του επιλέξιμου κόστος για τα πρότυπα η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί όμως να καλύψει την πλήρη χρηματοδότηση και για κάποιες μελέτες. Επίσης, σε περίπτωση που γίνεται στο πλαίσιο μιας μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας θα τη επιπλέον επιδότησης. Το πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας και στα σχέδια άμυνας και στα σχέδια ασφάλειας. Γιατί οι συμπολίτες μας περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή δέσμευση υπέρ της ασφάλειας και της άμυνας για να εγγυηθεί την απαραίτητη ασφάλεια σε έναν κόσμο που γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα ασταθής. Επίσης, οι πολίτες περιμένουν από μας περισσότερη συνεργασία για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι σε διεθνές επίπεδο, στο διεθνές προσκήνιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, να αφήσουμε να την ευκαιρία να κάνουμε πιο ανταγωνιστικό και καινοτόμο τον κλάδο μας, την αμυντική μας βιομηχανία που πραγματικά το χρειάζεται. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και δημοσιονομικά. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε να έχουμε τόσα πολεμικά αεροσκάφη, τόσα πολεμικά πλοία, γιατί έχουμε διπλάσιο αριθμό ναυπηγείων από τις Ηνωμένε Πολιτείε για υποτριπλάσιο ε, προϋπολογισμό. Ε, οπότε με το πρόγραμμα αυτό θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, θα κάνουμε κάποιες οικονομίες, αλλά θα ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας για να μην κατασπαταλούμε ε, την, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, με το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλουμε στην στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βελτιώσουμε την παρούσα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μια εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Γιατί στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την βιομηχανική και τεχνολογική βάση της ε, Ευρωπαϊκής Άμυνας. Και γι' αυτό λαμβάνουμε τέσσερις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Καταρχήν θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εταιρείε, οι δικαιούχε και οι υπεργολάβοι όντως ελέγχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι θέμα δηλαδή επιλεξιμότητας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το θέμα αυτό. Και το κριτήριο το 5% των Ευρωπαίων μετόχων που προτείνεται ε, είναι κάπως ασταθές κριτήριο και δυσεφάρμοστο και μάλιστα αδικαιολόγητο για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ε, το θέμα όμως του αποτελεσματικού ευρωπαϊκού ελέγχου είναι σημαντικό. Αυτή η έννοια του αποτελεσματικού ελέγχου είναι ήδη γνωστή και χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για τις αεροπορικές εταιρείε. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιος ε, ελέγχει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων της επιχείρησης και άρα να αναλύσουμε τον τρόπο διακυβέρνησης της επιχείρησης. Δεύτερη πρωτοβουλία ε, ε, αφορά το πότε αλλάζει ε, ο έλεγχος της επιχείρησης μετά από μια εξαγορά της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κρατημέλη θα πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα για να προασπίσουν την τεχνογνωσία και την τεχνολογία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τρίτον, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εντοπίσει τα προϊόντα και τις τεχνολογίες για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τρίτους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μειώσουμε την εξάρτησή μας. Τέταρτη συγκεκριμένη συνεργασία προάσπιση των αποτελεσμάτων των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα, ώστε να μην είναι προσβάσιμα για όλους. Με όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία μας στα θέματα τα αμυντικά. Θεωρώ σε ό,τι φορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ανεβέσει το θέμα ότι θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο είτε άμεσα είτε μέσω ε, μεγάλων ομήλων από τους οποίους θα αναλάβουν υπεργολαβίες. Προτείνω λοιπόν μια κατηγορία προγραμμάτων να αφιερωθεί ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τουλάχιστον 10% του συνολικού ποσού να διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι θεμελιώδες και για να εξασφαλίσουμε συμμετοχή όσο δυνατό μεγαλύτερη αριθμού κρατών μελών, αρκεί να είναι φυσικά εύρωστα και βιώσιμα τα σχέδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις από δύο διαφορετικά κράτη. Και αυτό το ελάχιστο κατόφλι είναι απαραίτητο ώστε να επιτρέψει πολυάριθμες συνεργασίες και τη χρηματοδότηση πολλών σχεδίων. Όσο το κατόφλι που αφορά τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις είναι υψηλό, τόσο περισσότερο θα θέσουμε σε κίνδυνο το πρόγραμμα και τα νέα βιομηχανικά σχέδια όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει αριστεία στο θέμα ασφάλειας και άμυνας μπορούν να αναλάβουν μέρος. Και αυτό το κριτήριο της αριστείας και της βιομηχανικής απόδοσης είναι ζωτικό κατά τη γνώμη μου. Επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπλακούν και ε, χρηματοδοτικά στις δράσεις του προγράμματος και γι' αυτό προτείνω μια ξεκάθαρη, ανεπιφύλακτη και γραπτή δέσμευση των κρατών μελών Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για την ασφάλεια και άμυνα μετά το 2020, αυτό θα εξαρτηθεί, ο προπολογισμό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματο. Γιατί καταλάβατε ότι για τη διετία 2019-2020 ε, θέτουμε τα θεμέλια αυτού του προγράμματος και αν πάνε όλα κατευχήν, στη συνέχεια θα προβλέψουμε συγκεκριμένα σχέδια που θα εγγυώνται την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Προσπάθησα να σας ενημερώσω και να συνοψίσω τη σημασία που έχει αυτό το ταμείο και ακριβώς επειδή έχουμε πολύ πιστικό χρονοδιάγραμμα καλό θα ήταν να, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να καταλήξουμε σε μία ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω οι συνάδελφοι κάπως να περιοριστούν στα σχολιά τους χρονικά σε ένα δίλεπτο. Λοιπόν, ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κ. Πόχε από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε, πολύ καλή. Έκανε προσπάθειες που τις εκτιμώ για τη βελτίωση του σχεδίου προτάσεως. Κοινό στόχο είναι το Ευρωπαϊκό, Ταμείο για την Άμυνα να πετύχει το στόχο του, να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να βελτιστοποιήσει τις δαπάνες των κρατών μελών. Είναι πιο λογικέ οι τροπολογίε τη εισηγήτρια. Γίνεται πιο λογικό το κείμενο και θα είναι ισχυρή η θέση του Κοινοβουλίου στον επικείμενο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Η έκθεση επικεντρώνεται επί της στατικής αυτονομίας της Ευρώπης. Καταρχάς, αυστηρή αιρεσιμότητα για εταιρείε που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα. Δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσει ότι θα συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα και αυτό είναι μεγάλο κενό. Δεν αναφέρεται τίποτα περί χρηματοδοτήσεως του προγράμματος. παρόλο που είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση θα είναι ένα επίμαχο ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες με στόχο το να δοθούν κίνητρα στα κράτη-μέλη και στη βιομηχανία να δημιουργηθούν κάποιοι όμιλοι, κάποια κονσόρσια στα οποία θα συμμετέχουν και εκπροσωπούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισαγάγει στα διαστημικά προγράμματα και στο μέτρο για την διασύνση της Ευρώπης περικοπές για την υποστήριξη του Ταμείου για την Άμυνα. Εγώ θα προτείνω μεγαλύτερη χρήση των ε, ποσών του προπολογισμού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης και ε, το θέμα της εξαγωγής των προϊόντων που σηματοδοτούνται. Λόγω της φύσεως των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο περιορισμών εξαγωγών. Όσον αφορά τις εθνικές νομοθεσίες και τον εθνικό έλεγχο, η αναφορά σε αυτά δεν αρκεί. Να υπενθυμίσω ότι στις 13 Νοεμβρίου εκπρόσωποι 23 κρατών μελών δεσμεύτηκαν να, έχουν συνεργασία στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφαλείας. Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική εντός ε, του Ευρωπαϊκού αυτού Ταμείου για την ε, Άμυνα. Και κάτι άλλο. Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτού είναι προς όφελος ε, των πολιτών μας, διότι η ασφάλεια είναι προς όφελος τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αυτό που δεν είναι προς όφελός μας είναι το να δίνουμε χρήματα σε κάποιες επιλεγμένες ε, εταιρείε που δεν δίνουν προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη και νομίζω ότι η θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι αρκετά στεναρή για να αποφύγει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι συμφωνείτε και υποστηρίζετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κρασνοντεύσκη. Ο κ. Κρασνοντεύσκη έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερος τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ο κλάδος αυτός, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι ε, πρόκειται να αναπτυχθεί ο κλάδος όταν έχουμε παρόμοιο δυναμικό σε όλες τι χώρες μέλη, όταν αξιοποιηθεί το δυναμικό και το ερευνητικό και το βιομηχανικό του συνόλου της Ευρώπης και όχι μόνο ενό τμήματο της Ευρώπης ή μερικών χωρών. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βιομηχανικές βάσεις και να γεφυρωθεί ε, το, η απόσταση μεταξύ αυτών των χωρών και την υπόλοιπο που δεν είχαν πρόσβαση μέχρι στιγμή σε διεθνή σχέδια. Ε, Δυστυχώ το σχέδιο έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη κάποιου ιστορικού παράγοντε, ιστορικά κριτήρια και τη διαφοροποίηση τη βιομηχανική βάση ε, στην Ευρώπη. Ούτε λαμβάνει δέντο υπόψη το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Επίση, ε, έχουμε διαφορετικέ δυνατότητε χρηματοδότηση. Και δυστυχώς ακόμη και οι τροπολογίε τη κυρίας Γκροστέτ παραλείπουν αυτά τα σημαντικά θέματα. Και χωρίς την χωρίς την λήψη υπόψη των δικών μας τροπολογιών, το πρόγραμμα ουσιαστικά θα ευνοήσει τις πολυεθνικές ήδη και θα ε, Αποβεί βάρο κάποιων ε, υφισταμένων ερευνητικών προγραμμάτων με εταίρου ή θα ευνοήσει μόλ, μόνο μερικούς βασικούς παίκτε της Ευρωπαϊκή Αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουν αρκετά σημεία στο κείμενο. Καταρχήν, στα κριτήρια για τη χρηματοδότηση θα πρέπει να προσθέσουμε ή να επιβραβεύσουμε ε, κάποιες νέες μορφές συνεργασίας, να προωθήσουμε νέες μορφές συνεργασίας Επίσης, ε, να λάβουμε όπως την ε, επιρροή της ε, συνεργασίας στην βελτίωση της τεχνολογικής βάσης και να λάβουμε υπόψη την ανάγκη συμμετοχής όλων των χωρών μελών στην ασφάλεια. Επίσης, να γίνει μια διαφοροποίηση των επιλέξιμων φορέων και δεν συμφωνώ με κάποιες δηλώσεις της εισηγήτριας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες ε, μέσες επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής ε, ε, είχαν στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας και το πρόγραμμα αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ, αλλά να τη συμπληρώσει. Θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, που είναι μια στρατιωτική συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε. Επίσης, ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε στο πρόγραμμα τη συμμετοχή και επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν και ε, χώρες ε, που συνεργάζονται με τρίτες χώρες. Να ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική ισορροπία που θα πρέπει να περιληφθεί στους δείκτες για την αξιολόγηση του προγράμματος. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ίσως ε, δεν προσέξατε ότι ε, ο χρόνος σας είναι της τάξης των δύο λεπτών και ε, χρησιμοποίησατε 6,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ όμως για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε, λέει ο κ. Κράσινοντέμψικη. Εκπρόσωπος της ομάδας των φιλελευθέρων Άλντε, ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Συγήτρια για την ποιοτική εργασία της καθώς και για την συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φαίνεται να φτάνει στο κατάλληλο χρονικό σημείο σε ό,τι αφορά και την κυριαρχία και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής άμυνας. Και χρειάζεται πράγματι μια συνολική βελτίωση της διευρωπαϊκής συνεργασίας. Υποστηρίζω τις απόψεις που εκφράζει η εισηγητρία σε μεγάλο βαθμό και πολλές από τις προτάσεις της. Ωστόσο, ορισμένα σημεία θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Πρώτα, πράγματι, ο αποτελεσματικό έλεγχος από την Ευρώπη, από τους Ευρωπαίους των επιχειρήσεων, είναι δύσκολο για τους μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Είναι ένα πρώτο θέμα λοιπόν αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι η πηγή των χρηματοδοτήσεων, η προέλευση των χρηματοδοτήσεων. Θα είναι ενδιαφέρον να συζητηθεί αυτό. Θα είναι επιθυμητό να σημειωθούν τα συγκεκριμένα νούμερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το καθεστώς τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ω χρηματοδοτικού οργάνου θα πρέπει να τροποποιηθεί για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα τη άμυνα. Θα πρέπει να είναι κανεί πάρα πολύ αυστηρό ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε. Χωρί να έλθουμε σε αντίθεση με του συμμάχου μα ιδίω βέβαια τη Ατλαντική Συμμαχία, αλλά άλλο θέμα είναι να αυξήσουμε τη, βάση, τη βιομηχανική μας βάση, εάν δεν είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας στο διεθνές επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηριχθεί και θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ανάγκες αυτές από το προσεχές ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο εκπρόσωπος της ομάδας των Πράσινων, κύριος Μπιουτικόφερ στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Δεν ε, μας αρέσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν ε, προχωρεί αρκετά. Ο σκοπός του όλου θα πρέπει να είναι να μειωθούν οι περιττές δαπάνες, να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών μας και να αυξηθεί και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όπως είπε και ο συνάδελφος μου προηγουμένως. Όμως δεν σημαίνει αυτό. Η συζήτηση που διεξάγουμε τώρα εδώ οδηγεί μάλιστα σε ακόμα πιο αρνητική κατεύθυνση. Οι συνάδελφοί μου μιλούν για γεωγραφική ισορροπία, αυτό όμως ε, δεν έχει καθόλου σχέση με την αποτελεσματικότητα. Στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ούτε αυτό πρέπει να αποτελεί κίνητρο. Συμμετοχή του μέγιστου αριθμού των χωρών μελών, ούτε αυτό είναι κριτήριο αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας. Αυτά που λένε οι συνάδελφοι είναι να ξεκινήσουμε ένα νέο γύρο επιδοτήσεων στον αμυντικό τομέα χωρίς να επιμείνουμε σε αυτά όπου θα πρέπει να επιμείνουμε, δηλαδή περισσότερη απόδοση των επενδύσεών μας, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερες σπατάλες. Οι χώρες μέλη δαπανούν σήμερα τα τριπλάσια χρήματα για άμυνα από ό,τι η ρωσική κοινοπολιτεία, χωρίς να βρίσκονται σε θέση να μπορούν να ορθώσουν το παραστημά τους απέναντι στη ρωσική κοινοπολιτεία, για παράδειγμα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να κοιτάξουμε στα μάτια της πραγματικότητας. Δεν μιλούμε εδώ για πολιτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλούμε για στερέωση, σταθεροποίηση μιας ολόκληρης βιομηχανίας. Αν δεν το κάνουμε σωστά, ας το αφήσουμε το εγχείρημα αυτό. Δεύτερο, από πού έρχονται τα χρήματα. Περικόπτουμε δαπάνες που δεν θα πρέπει να περικόπτονται και δεν επιμένουμε ως χώρες μέλη να τοποθετήσουν τα χρήματα εκεί όπου θα πρέπει, αν πράγματι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα αυτό. Και τρίτο, η δομή δίνει υπερβολικό λόγο στη βιομηχανία σχετικά με το πού θα γίνουν οι χρηματοδοτήσεις, που θα γίνουν οι επενδύσεις. Αυτό είναι αμφι, αμφισβητήσιμης αξίας. Όχι μόνο δηλαδή σπαταλούμε χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με αποδοτικότερο τρόπο, επιτρέπουμε μάλιστα στην βιομηχανία να συναποφασίζει για το πού θα σπαταλήσουμε τα λεφτά αυτά. Θεωρώ ότι είναι απολύτως αποπροσανατολισμένη η προσπάθεια αυτή να πατήσουμε γερά τα φρένα και να ξεκινήσουμε προς άλλη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας, λέει ο πρόεδρος Κόχλιτσεκ. Θα ακολουθήσει τώρα ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Αριστεράς, κ. Σιλικιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμενας αποτελεί κατά την άποψή μα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για οικοδόμηση της Στρατιωτικής Ένωσης. Αυτή είναι και ουσία και δυστυχώς πρέπει να πω ότι και μέσα από την έκθεση της συναδέλφους που εκτιμώ τη δουλειά της παρόλο που σε πολλά σημεία διαφωνώ της ε, Κροσέτε ε, γίνεται αποδεκτό αυτό το πράγμα. Κατατέθηκε μια πρόταση από την Κομισιό χωρίς καν εκτίμηση των επιπτώσεων με τη δικαιολογία του κατεπήγοντος και ζητείται να γίνουν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία ώστε η Ένωση να αποτελέσει ισχυρότερο τέρο στον στρατικό τομέα. Και μάλιστα όπω αναφέρθηκε και εδώ, προ επίτευξη αυτού του στόχου μέσα σε δύο χρόνια ζητείται να δοθούν 500 εκατομμύρια μονάχα από την Κομισιόν, ενώ το υπόλοιπο 80% του συνολικού κόστου εν καιρό κρίση θα καλεστούν να πληρώσουν τα κράτη-μέλη. Αφού θεωρείται ότι υπάρχει ένα τότε μεγάλο κοντίτι διαθέσιμο, γιατί δεν το αξιοποιεί η Ένωση για την πρόθεση τη επαναβιομηχανοποίηση ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη ε, στα κράτη-μέλη του Νότου που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τι πολιτικέ λιτότητα. Γιατί δεν κατατέθηκε μέχρι σήμερα η πρόταση για ανάπτυξη μια ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική, η οποία να αντιμετωπίσει την ανεργία και να συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και στη ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των λαών, και αντί τούτου μιλούμε για ενίσχυση τη αμυντική βιομηχανία. Τα 500 εκατομμύρια που θα διαδέσει η Κομισιόν Όπω αναφέρθηκε και από τον προλαλήσαντα, το συνάδελφο από του πράσινου, θα αποκοπούν από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκαλώντα έτσι διπλή ζημιά. Για παράδειγμα, τη στιγμή που γίνεται συζήτηση για την άγκη ενίσχυση του προγράμματο συνδέοντα την Ευρώπη, καθώ κράτη και περιοχέ τη Ένωση βρίσκονται ακόμα ε, απομονωμένε από τα δίχτυα, προτείνεται να αποκοπούν 145 εκατομμύρια για να επενδυθούν στην αμυντική βιομηχανία. Εμείς το αυτό το θεωρούμε και λαθασμένο και απαραδεκτό. Το άρθρο 41 παράγραφος 2 τη Συνθήκη τη Ένωση, αναφέρει ξεκάθαρα πω οι δαπάνε που προκύπτουν από επιχειρήσει που έχουν στρατιωτικέ ή αμυντικέ συνέπειε δεν πρέπει να χρεώνονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Και όμω δυστυχώ, αυτό είναι που επιχειρείται σήμερα με τη δικαιολογία του άρθρου 173 για την βιομηχανική πολιτική. Α είμαστε ειλικρινεί, στην τελική αυτό που προτείνεται είναι να αποκοπούν λεφτά από αναπτυξιακέ πολιτικέ για να επενδυθούν στην ενίσχυση αμυντικών και στρατιωτικών δομών τη Ένωση. Εμεί θεωρούμε ότι θα καταθέσουμε τροπολογίε. Βεβαίω, όσε τροπολογίε και να καταθέσουμε, η ουσία αυτή καθ' αυτή δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό το λέω ξεκάθαρα από την αρχή ότι η δική μα ομάδα, η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, θα απορρίψουμε συνολικά αυτή την πρόταση για αυτή, γιατί αυτή η θέση κατά την άποψή μας είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει εκπρόσωπος από την ομάδα EFDD, από την ομάδα ENF. Καλά. Άρα Κάποιος διακόπτει από κάτω. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει την εισηγήτρια, έτσι δεν είναι. Είναι σαφές ποιος είναι ο εισηγητής, έτσι δεν είναι. Βεβαίως θα λάβετε το λόγο κύριε Έλερ. Στο δεύτερο γύρο. Έτσι είναι ο κανόνας. Minuten, Πόσα λεπτά έχω κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Σούλτσε πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της που τη βρίσκω σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη, περιέχει πολλά θετικά πράγματα. Ένα πολύ θετικό μου φαίνεται το 20% οροφή σε αυτά τα περιορισμένα χρηματοδοτικά κονδύλια των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση πρωτοτύπων. Ωστόσο έχω και μια κριτική παρατήρηση που θα ήθελα να θέσω υποσυζήτηση. Είναι η προσέγγιση που λέει ότι στην έρευνα θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο εταιρείε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζονται μηχανισμοί προστασία, ασφάλεια κλπ. για τι πληροφορίε, αλλά είναι νομίζω λάθο ε, να υπερπεριορίσουμε τα πράγματα. Μπορεί να φοβηθεί κανεί ότι κάποιο know-how θα διαρρεύσει, αλλά το αντίθετο επίσης είναι σωστό ότι μπορεί και να εισρεύσει κάποιο know-how από άλλες χώρες προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ίσως ναι, καταρχήν μεν οι χώρες μέλη του ε, ΝΑΤΟ που θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και δεύτερο αμοιβαιότητα. Για παράδειγμα, τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται για αμυντικά θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζουν σχετικά σημαντικό ρόλο στην έρευνά μας και εμείς στη δική τους έχουμε για παράδειγμα καλή συνεργασία με χώρες όπως η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη. Αυτές να μπορούν να συμμετέχουν. Νομίζω λοιπόν ότι κάπως ε, διανοητικά πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ. Βεβαίω αντιλαμβάνεστε ότι σε περίοδο συνόδου τη Ολομέλεια δεν θα μπορούσα να σα δώσω τόσο πολύ χρόνο. Ο κύριο Χακμάρκ είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ένα βασικό σημείο θα να τονίσω. Ότι η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα τα καλύτερα δυνατά συστήματα και όπλα για την πράσπιση των κοινωνιών μας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη έρευνα, την καλύτερη καινοτομία, τις καλύτερες γνώσεις και δεξιότητες από όπου και να προέρχονται, να βρίσκονται όμως στην Ευρώπη. Είναι πιο σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα, τη δυναμικότητα για να αναπτύσσουμε τεχνολογία εχμής στην Ευρώπη αντί να συζητούμε πού θα παράγεται στην Ευρώπη το κάθε κομμάτι. Είναι καλό να έχουμε διεθνείς φορείς που θα συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικού και δυναμικότητας στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα και το κράτησα στο ένα λεπτό. Ευχαριστώ υπέροχα, λέει ο Πρόεδρος. Συνάδελφε Κοντουσόφσκι, έχετε το λόγο. Κύριε Κοσινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος και θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει πόρους, αλλά δεν συμφωνώ ότι 150 εκατομμύρια ευρώ, που το είναι το 1 τρίτο του συνολικού ποσού, ε, το πήραν από τα διαστημικά προγράμματα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Επίσης, ανησυχώ και για κάτι άλλο. Για το πρόγραμμα Γαλιλαίος που βρίσκεται στην τελική του φάση και φοβούμε ότι Αργότερα θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε να βρούμε χρήματα για τη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου, που πάντα ίσχυε αυτό. Πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε χρήματα για το Γαλιλαίο. Αναφέρθηκε η συγγήτρια στην ανάγκη σύμπραξη μεταξύ διαστημική πολιτική και αμυντική πολιτική. Κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει και σε αυτό το πρόγραμμα να το λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει τα διάφορα διαστημικά προγράμματα να συμπεριληφθούν. Δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν τα προγράμματα αυτά για να προχωρήσουμε στον άλλο τομέα. Τον αμυντικό, ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Συμφωνούμε νομίζω. Όχι μόνο δύο-τρεις ομιλητές, μεταξύ μας συμφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, από άλλους πόρους να εξευρεθεί η χρηματοδότηση. Όχι από τρέχοντα προγράμματα όπως είναι το Γαλιλαίος και άλλα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας διότι σχεδόν όλοι είπαν το ίδιο πράγμα. Τη χρηματοδότηση ανέφεραν. Επόμενος, ο κ. Έλερ, παρακαλώ, συνάδελφοι, συνάδελφοι, θα, θα, είστε, θα, είστε σύντομος, θα είμαι αυστηρός μαζί σας και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά μπορείτε να μιλήσετε λίγο παραπάνω. Ε, ήθελα αρχικά να συμφωνήσω με τον κύριο Μπιουτικόφερ, αλλά κάτι τέτοιο δεν βελτιώνει τη συζήτηση. Στην έκθεση της κυρίας Κροστέτ αναφέρεται περί τίνος πρόκειται. Λίγο πολύ δίνουμε συνέχεια στα όσα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Δεν αποφάσισε μόνο του το Συμβούλιο την γεωγραφική ισορροπία. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι έχουμε μια συνολική στρατηγική ως Ευρωπαίοι βρισκόμαστε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς σχετικά με την Ατλαντική Συμμαχία, με τη Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πρέπει να υλοποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει και το πρόβλημα της χρηματοδοτήσεως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θεσπίσουμε νέες πολιτικές με τα μισά χρήματα. Διότι υπάρχει και το πρόβλημα ότι καν δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και το 2022 κινδυνεύουμε να μην έχουμε πλέον χρηματοδότηση. Και απλώ θα έχουμε ανοίξει το κενό ανάμεσα σε υποχρώσεις και πληρωμές. Το δεύτερο είναι η ίδια φύση του πράγματος. Η ίδια η πρόταση είναι σχετικά ασαφής. Όταν βλέπω τις δημοσιονομικές ρυθμίσεις, τι γίνεται για το IP management ας πούμε ή το σύστημα κατανομών, είναι αρκετά εκπληκτικό ότι ένα κοινοβούλιο δέχεται να κάνει τέτοια πράγματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον επίγοντα χαρακτήρα, αλλά κανονικά τα πράγματα αυτά θα έπρεπε να βασίζονται πάνω σε δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι ασαφής τα πράγματα αυτά και στην ουσία σημαίνουν μια προκαταβολή κεφαλαίου εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη γεωγραφική κατανομή. Έχει σχέση το πού βρίσκεται, πού ξεκινά το πρόγραμμα. Και θα πρέπει να γίνει να γίνουν προτάσεις ώστε να ωφεληθούν όλες οι χώρες μέλη. Όμως είναι σαφές ότι θα ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε χρήματα σε κάποιους οι οποίοι θα πούν μετά «Όχι, δεν θέλουμε χρήματα για τη βιομηχανία μας». Χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και όχι να φτάσει να καταλήξει να είναι επιδότηση βιομηχανίας. Το άλλο θέμα που κάπως με τρομάζει είναι ο προσανατολισμός. Τα χρήματα φαίνονται πολλά. Καταρχήν το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τη στόχευση να μην ανταποκριθούμε απλά σε ένα ευχολόγιο της βιομηχανίας. Θα πρέπει να δούμε τι λέει και στο προήμιο εδώ, δηλαδή κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν πρόκειται απλώς για ενίσχυση κάποιων εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας σε δύο-τρία συστήματα και για να καθησυχάσω τους συναδέλφους 80% των χρημάτων προέρχεται από τις χώρες μέλη. Επομένως οι χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν και ισχυρά κίνητρα για να το κάνουν. Και κάτι που δεν μπορεί να επιλύσει το πρόγραμμα είναι όποιος δεν επιθυμεί από τις χώρες μέλη να χρηματοδοτήσει, δεν πρόκειται και να λάβει χρήματα για τη βιομηχανία του. Δεν είναι δηλαδή δωρεάν η συμμετοχή. Είναι μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα προς τις χώρες μέλη, ώστε να καταβάλουν κοινέ προσπάθειες για προώθηση τεχνολογίας, για κοινή συμμετοχή σε συστήματα αμυντικά και άλλα και όχι απλώς ένα ανοιχτό πρόγραμμα επιδότησης βιομηχανίας. Αυτά τα πράγματα, παρόλη την σχετική κριτική, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να τα προωθήσουμε και να αποδώσει η προσπάθεια αυτή. Διότι εγκρίνουμε κάποια global strategy και μετά φέρνουμε τόσα πολλά αντίθετα επιχειρήματα για την πρώτη δόση αυτή των 500 εκατομμυρίων που τελικώς δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μετά από μια πρώτη φάση θα δούμε κατά πόσον θα πρέπει να προχωρήσουμε και πώς. Αλλά θα πρέπει να δεχθεί καθαρά ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχθεί ως σχεδιασμό για χρηματοδότηση από τον παρόντα κοινοτικό προϋπολογισμό, διότι αυτό δεν αρκεί. Ευχαριστώ κύριε Σάδεφε. Νομίζω ειδικώ αυτό που είπατε για το ευχολόγιο της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας είναι σημαντικό γιατί θίγει πολλές χώρες. Επόμενος ο μιλητής ε, στον κατάλογο είναι ο η κυρία Ντελάγκε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ε, μία από τις βασικές εκθέσεις ε, που θα πρέπει να προωθήσει η κυρία Γκροστέτ και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Δύο είναι τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Το θέμα του ελέγχου και το θέμα τη ε, ιδιοκτησία, τη πνευματική ιδιοκτησία, για παράδειγμα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε, αυτό είναι το πρώτο σημαντικό θέμα. Και δεύτερο, ε, αυτό, αυτή η μαγική συνταγή, τουλάχιστον τρει επιχειρήσει ε, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Εγώ κατάγομαι από μια σχετικά μικρή χώρα και ε, θεωρώ σαφέ ότι αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση θα λειτουργήσει αν όλοι έχουν την αίσθηση ότι κάτι κερδίζουν. Γιατί λοιπόν κάποιες χώρες ε, ε προτιμούν να αγοράσουν ε, αμερικανικά μαχητικά ε, γιατί ε, προτιμούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη βιδών και άλλων ανταλλακτικών από το να πρέπει να κατασκευάσουν ίδιες μαχητικά. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την αμερικανική τεχνολογία και να κατασκευάσουμε τα δικά μας μαχητικά και γι' αυτό θέλουμε όλες το δυνατό περισσότερες χώρες που να συμμετέχουν. Και όσο περισσότερες χώρε συμβάλλουν, τόσο θα είναι και η πολιτική υποστήριξη σε πολιτικό επίπεδο για τέτοιου είδου προγράμματα στα κράτη-μέλη. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτή τη μαγική φόρμουλα των τριών επιχειρήσεων και δύο κρατών να πούμε ότι για, ένα επιπλέον, για κάθε επιπλέον κάθε ε, για, ένα, για κάθε επιπλέον κράτος που θα συμμετέχει να αυξάνουμε κατά ένα ποσοστό τη χρηματοδότηση για να είναι ε, δεν είναι αρκετή κίνητρο για τα κράτη να συμμετέχουν και επίσης να δούμε από πού θα προέρθουν τα υπόλοιπα κονδύλια. Σας ευχαριστώ. Βλέπετε κυρία, ε, κυρία α, Λάγκε, παρόλο που κανονικά δικαιώσατε ένα λεπτό, σας έδωσα δύο. Η κυρία Μούντι, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια, ε, την κυρία Γκροστέτ, ε, για την εξαιρετική της προσπάθεια δεν θα επαναλάβω τα σχόλια των συναδέλφων. Πάντως, αν θέλουμε πραγματικά να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα πρέπει να λάβουμε κυρίως υπόψη δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή τι θα καταστήσει πραγματικά αποτελεσματικό το πρόγραμμα, τι θα αποφέρει οι καρπούς και όπως είπαν οι συνάδελφοι, όσο περισσότερους περιορισμούς έχουμε και φραγμούς, τότε θα το αντισταθμίσουμε, πρέπει να το αντισταθμίσουμε με την αποτελεσματικότητα. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα, ένα ζήτημα που μας καίει αυτή τη στιγμή, θα επηρεάσει και το χρονοδιάγραμμα τα αποτελέσματα, αν συμπεριλάβουμε σημαντικούς περιορισμούς. Επίσης, συμφωνώ με τους συναδέλφους και τα σχόλιά τους για το προϋπολογισμό. Ε, δεν θέλω να κλέβουμε από τις τσέπες άλλων προγραμμάτων για να τροφοδοτήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να αποφύγουμε ό,τι συνέβη σε άλλα προγράμματα, σε ρίχνωσή τους υπέρ ε, τρίτων προγραμμάτων και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, να αντισταθούμε σε περικοπή άλλων προγραμμάτων για να το χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο. Κυρία Βέρνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Γκροστέτ για την έκθεσή της. Οφείλω να ομολογήσω ότι παρά τη θετική εντύπωση που δημιουργήθηκε για την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ δεν συμφωνώ μαζί της. Εμείς οι βουλευτές της S5 πάντοτε στηρίξαμε την εξέλιξη αυτή και βεβαίω και στα πλαίσια τη διαφρομένης συνεργασία η οποία εγκρίθηκε μόλι προλίγων μόλις προ λίγων εβδομάδων ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Υπάρχουν πράγματι αυτέ οι διπλέ ε, ε, δομές, οι επικαλύψει. Μπορούν τα χρήματα και πρέπει να διατεθούν με αποδοτικότερο τρόπο. Και υπάρχουν και μελέτε που δείχνουν ότι η αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονομήσει πολλών δισεκατομμυρίων και 2-3 δισεκατομμυρίων. Και το pooling και sharing σε ό,τι αφορά τις ικανότητες, λέμε ναι επίσης στην κατάργηση των γραφειοκρατικών εμποδίων, αλλά βάζω ένα σημαντικό ερωτηματικό για την διάθεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με τον τρόπο που προτείνεται. Μία σύντομη παρατήρηση. Το άρθρο 173. Εδώ λείπει μια καθαρή ρύθμιση για ποια έργα μπορούν να διατίθεται τα χρήματα δίνουμε 1,5 δισεκατομμύριο χωρίς να συναποφασίζουμε. Και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ανάληψη, την ανάληψη κονδυλίων από πόρους όπως ο, αυτό που διατίθεται για τον Γαλιλαίο για να δοθούν στην αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. καθυστερήσαμε λίγο και με τη δική σας ομιλία. Η κυρία Αλιό Μαρή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και κάποια χρόνια δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και έχω κάποια σχόλια να κάνω. Πρώτα απ' όλα τη χρηματοδότηση. Πράγματι αυτά τα 100 δισεκατομμύρια είναι λίγα, αλλά για τη συμμετοχή των κρατών. Πρέπει να δώσουμε κάποια κάποια κίνητρα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια κατανομή χρημάτων υπό τον όρο ότι και οι χώρες θα συμμετέχουν και με ένα σημαντικό τρόπο, ακόμα και πιο μικρές χώρες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, να υπενθυμίσω σε κάποιους ότι αν, δούμε, αν πάρουμε χρήματα από άλλους προϋπολογισμούς, η αμυντική βιομηχανία αφορά εκατοντάδες θέσεις, χιλιάδες θέσεις ε, απασχόλησης, πάρα πολλές επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει και διτή έρευνα που λαμβάνει η χώρα στον τομέα της άμυνας, αλλά μια έρευνα που έχει και αποτελέσματα και συνέπειες και χρήσεις και στον τομέα τον πολιτικό. Αναφέρατε κάποιοι το Γαλιλαίος. Στο Γαλιλαίος, στο πρόγραμμα Γαλιλαίος υπάρχει ένα τμήμα που αφορά την αμυντική χρήση. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε δυνατότητα την τεχνολογική, την τεχνογνωσία και το προσωπικό για να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας της αμυντικής. Αρκεί να δείτε τι έχει δημιουργηθεί. Το Ραφάλ, το Tiger και άλλα ε, οπλικά συστήματα και βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα χωρίς να χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα να προσφεύγουμε σε συμμαχίες με άλλες χώρες που αυτό δημιουργεί και κάποιο βαθμό εξάρτησης. Ευχαριστώ. Το ίδιο σχόλιο έχω, όπως το προηγούμενο. Και τώρα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας παρακαλώ, τρία λεπτά. Μόνο τρία λεπτά να είναι η συνεισφορά σας στη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Θα επιμείνω επί τριών σημείων που εθίγησαν Καταρχάς, όσον αφορά τους δικαιούχους, στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι δικαιούχοι και η ανταγωνιστικότητα αυτό αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Γι' αυτό προτείναμε ένα κονδύλι αρκετά περιορισμένο ε, και γραμμή αυστηρή όσον αφορά τους δικαιούχους. Τα κριτήρια του 50% είναι μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατανοούμε ε, και ότι χρειάζεται μια προσέγγιση για το αποτελεσματικό έλεγχο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και από αυτή τη βάση. Δεύτερο, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λοιπόν, στόχος δεν απλώς να ευνοήσουμε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να δρομολογήσουμε προγράμματα που θα είναι υποφελή για όλες τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένες και τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τούτο λεχθέντος, η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνει βάση αριστείας, βάση διαγωνισμών και βέβαια οι επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προτείνουν διάφορα προγράμματα. Αν τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις προτείνουν καλά προγράμματα που θα επιλεχθούν βάση αριστείας, τότε όλοι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά. Όσον αφορά ειδικέ διατάξει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί για μια βελτίωση σχετική του κειμένου. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα σημείο που είναι σημαντικότατο και για το Συμβούλιο. Άρα είμαστε απολύτως ανοιχτοί προς βελτίωση αυτού του τμήματος του κειμένου. Τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις σχέσεις με το διάστημα. Όπως ξέρετε είναι κάπως δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα θεσμικό όργανο, μας λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά τα χρήματα από ε, μεταφορά και άλλοι που μας λένε αποκλειστικά νέους πόρους που να χρησιμοποιείται. Η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπου στη μέση, αλλά βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα δύο θεσμικά όργανα ώστε να βρεθεί μια λύση ε, που να ταιριάζει. Τούτου λεχθέντος όσον αφορά το διάστημα θα επέμενε επί το εξή. Τα αμυντικά προγράμματα μπορούν να αφελούν σε όλους τους τομείς. Και βεβαίως ε, και κυρίως το διάστημα. Η σχέση μεταξύ διαστήματος και άμυνας γίνεται ε, όλο πιο στενή και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του διαστήματος θα μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτά τα προγράμματα βεβαίως αν υποβάλλουν σχετικά σχέδια προγραμμάτων που θα εξεταστούν με μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Ήρθε και πάλι η ώρα σας κυρία Γκροστέτ. Μπορείτε να συνοψίσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και το μήνυμά τους ελήφθη, οι παρατηρήσεις τους έχουν καταγραφεί και θα προσπαθήσω να συνδυάσω ε, στην απάντησή μου τα θέματα τα πιο σημαντικά προς συζήτηση. Για τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 500 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία. Και φυσικά τα κράτη-μέλη, όπως πολύ εύστοχα είπε η κυρία Λεωμαρή, θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτά. Για το 2019-2020 είναι 2 δισεκατομμύρια που θα πρέπει να συμβάλλουν τα κράτη-μέλη στα 500, ε, εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και φυσικά χρειάζεται ωραία, καλά, αξιόλογα προγράμματα για να χρηματοδοτηθούν και αντιλαμβάνομαι ότι φοβάστε μην ε, μονοπολίσουν μερικά κρατημέλη μόνο τη χρηματοδότηση. Όχι, θα ήθελα να σας καθησυχάσω, γιατί αυτό που προέχει και θα ληφθεί υπόψη είναι η ποιότητα των σχεδίων. Και κάθε κράτος θα μπορεί να ε, προτείνει σχέδια συμβάλλοντας φυσικά στη χρηματοδότησή τους. Και επίσης μιλούμε για συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Δεν πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που θα υποκαταστήσουν τα σχέδια που έχουν ήδη ε, τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο για την άμυνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γνωρίζω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει θέση. Είναι ήδη δεδηλωμένη η πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών που δεν θέλει ούτε κουβέντα για ε, μεταφορά κονδυλίων από υπάρχοντα προγράμματα. Θα πρέπει όμως να βρούμε μια ισορροπία στην πρόταση χρηματοδότησης. Όντως κάποιες δημοσιονομικές γραμμές ίσως χρησιμοποιηθούν ακριβώς γιατί είναι συμπληρωματικέ και ακριβώς γιατί αφορούν ε, και το πολιτικό σκέλος ή αφορούν θέματα διαστήματος και έχουμε και τα περιθώρια. Περιμένω να διαμορφωθούν οι διάφορες θέσεις και ξέρω ότι η πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα είναι αρκετά μονοσήμαντη. Θα πρέπει όμως μετά να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις mid-cap, φυσικά ε, και αυτές τις περιβάλλουμε, περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμα και καλούνται να λάβουν μέρος. Και από αυτές εξαρτάται. Πιστεύω όμως ότι το γεωγραφικό κριτήριο δεν είναι εύστοχο το, τα κριτήρια θα πρέπει να αφορούν περισσότερο την αριστεία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των προτάσεων. Μακάρι να εμπλακούν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν ευχή έργων και απαραίτητο για την επιτυχία του συνολικού προγράμματος. Αλλά γνωρίζω ότι κάποιες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, στα κράτη-μέλη είναι πιο πρόσφορες, ε, πιο δεκτικές σε τέτοια προγράμματα. Γιατί έχουν πλούσια πείρα και μεγάλη ανταγωνιστικότητα, οπότε θα είχαν και μεγαλύτερη ε, ροπή προς τέτοια προγράμματα και σχέδια. Επίσης, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, το ζητούμενο εδώ είναι η αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα είναι η ουσία αυτού του προγράμματος. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για το θέμα αυτό της αποτελεσματικότητας. Θέλουμε να εδραιώσουμε αυτή τη βιομηχανία, την αμυντική βιομηχανία που πρέπει να είναι ιδιαίτερος καινοτόμα και ενατεριστική και γι' αυτό και πιο αποτελεσματική. Προσπαθώ εδώ να συνοψίσω. Μας λέτε να μην γίνουμε Άγιοι να μην λάβουμε υπόψη όλα τα, όλες τις επιθυμίες και φυσικά θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας για την πρώτη φάση του 2019 και 2020, το είπα, και στην αρχική μου παρατήρηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποιες είναι οι προτεραιότητες και πού μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, ε, ε, θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Σιλικιώτη που είπε να μην περικόψουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Όχι, που δεν είναι, δεν πρόκειται να θίξουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα να τον καθησυχάσω και να τον διαβεβαιώσω. Νομίζω ότι κάλυψα τα ουσιώδη γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι μίλησαν για τα ίδια θέματα. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας, ε, συνάδελφοι, και περιμένω και τις τροπολογίες σας. Για να βελτιώσουμε το κείμενο της έκθεσης. Είμαι απόλυτα δεκτική και στη διάθεσή σας. Θέλω να συζητήσουμε με βάση τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Θέλω πάντως, και αυτό είναι το βασικό να έχουμε μια ισχυρή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δείξουμε πυγμή απέναντι στο Συμβούλιο. Γιατί σίγουρα θα υπάρχει διάσταση απόψε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν όμω έχουμε ισχυρή θέση διαμορφωμένη μεταξύ μα, θα έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στο Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Γκροστέτ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή πολλές και διάφορες παρατηρήσεις. Καταρχήν, διορία για την κατάθεση τροπολογιών. 30 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία. 30 Νοεμβρίου 2017, 12 το μεσημέρι, λίγη διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Εξέταση των τροπολογιών. 11 Ιανουαρίου 2018. Δημόσια ακρόαση. 22 Ιανουαρίου 2018 ψηφοφορία στην Ήτρε. Μάλλον στις 21 Φεβρουαρίου του χρόνου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ανάλογα με το αν θα καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Άλλα σχόλια υπάρχουν για τα σημεία της ημέρησης διάταξης της απογευματινής. Όχι. Οπότε αύριο, ημέρα Τρίτη, 28 Νοεμβρίου. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 9 το πρωί και κλεισμένα των θυρών. Θα είναι η συνεδρίαση των συντονιστών και στις 10 θα ξεκινήσουμε τη δημόσια συνεδρίαση με τις ψηφοφορίες ενός ογκοδέστατου πακέτου ε, ψηφοφοριών. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.